<clears throat> Bien, mesdames et messieurs, chers collègues. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση που σήμερα θα αφιερώσουμε στη βιομηχανία της ασφάλειας στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα που το αναφέρουμε συχνά, αλλά όχι με τους άμεσα ενδιαφερόμενους δυστυχώς. Και έχουμε πολλές πολιτικές προσωπικότητες ε, και θεσμικούς παράγοντες. Είχαμε πρόσφατα τους επιτρόπους Γιάννη και Μπαρνιέ, φυσικά και εκπροσώπους της ΕΙΕΔ ή εκπροσώπους των ε, χωρών μελών που μας επισκέπτονται και που μας εκθέτουν τις απόψεις τους για το τι περιμένουν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου που θα αφιερωθεί στην άμυνα, αλλά δυστυχώς ε, ελάχιστα καθόλου μέχρι στιγμής δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τους ίδιους τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, του ίδιου του κλάδου. Και λογικό είναι να δώσουμε και σε αυτούς την ευκαιρία να εκφέρουν τη γνώμη τους, γιατί μιλούμε για μια πολύ σημαντική φάση της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Μιλούμε για το, τις δυνατότητες μας, τις θετικές μας ικανότητες, ε, για πολλά σχέδια που υπάρχουν, αλλά να ακούσουμε και τη φωνή των βιομηχάνων, των εκπροσώπων του κλάδου. Γι' αυτό και διοργανώσαμε σήμερα τη δημόσια ακρόαση, στην οποία θα συμπεριληφθούν και κάποια θέματα που δεν είχαμε προβλέψει κατά τη στιγμή της διοργάνωσης. Για παράδειγμα, συζητήσεις σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί διαβάζοντας ε, την διαπραγματευτική εντολή με τη μορφή που έχει σήμερα, ε, φαίνεται ότι καλύπτει και τη, τη βιομηχανία ασφάλεια και άμυνα. Και μάλιστα το συζητήσαμε αυτό και στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Σω ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και σήμερα. Επίση, έχουμε τη Γαλλική Λευκή Βίβλο που δημοσιεύθηκε και ο, ο Γάλλος Υπουργό Άμυνα ε, ήρθε στην κοινή συνεδρίαση τη Επιτροπή ε, Εξωτερικών και Επιτροπή Άμυνα την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία την Παρασκευή μίλησε για την εθνική άμυνα. Ε, αναφέρθηκε στις ε, αδυναμίες και τα κενά που υπάρχουν στην Ευρώπη στο επίπεδο αυτό. Οπότε το θέμα των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων της ε, στρατιωτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό. Και ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους μας που μας έκαναν την τιμή να έρθουν σήμερα. Ε, Πολλοί δε μερικοί ε, είχαν, βρήκαν χρόνο να περάσουν και από τις Βρυξέλλες, ενώ είχαν αλλού Ευχαριστώ τον κύριο Ταραπιά που είναι ο πρόεδρο άμυνα τη ΑΕΣΤΕ και γενικό διευθυντή τη ΔΑΣΟ, ο Ντανιέλ Ρόμιτι που είναι διευθυντή τη Αγκούστα Westland και τον κύριο Γιάν Πι, ή ε, που είναι γενικό διευθυντή τη ε, Σουηδική Βιομηχανία, ε, τη Ένωση μάλλον Βιομηχανιών Ασφάλεια και Άμυνα. Επίση έχουμε και τον Κριστιαν Μέλινγκ από το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα διεθνή θέματα και θέματα ασφάλειας. Ο κύριος Μέλινγκ μάλιστα εκπονήθηκε τη στιγμή μία μελέτη ε, μετά από αίτημα τη υποεπιτροπή ε, μα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Να προσθέσω και τον συνάδελφο Μίκαελ Γκάλερ, που είναι παρόν και θα συντάξει και έκθεση πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Βιομηχανική και Αμυντική Βάση. Πολύ σημαντική έκθεση πρωτοβουλία που θα εξεταστεί στι ε, επιτροπέ ε, βιομηχανία, εσωτερική αγορά και απασχόληση που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενε και αρμόδιες για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Τραπιέ, τον κύριο Ρομίτη και τον κύριο Πιέ. Θα έχουμε μια, ένα χρόνο για ερωταπαντήσεις, κατόπιν στον κύριο Μέλινγκ και μετά πάλι θα ακούσουμε τους καλεσμένους μας για τα συμπεράσματα. Έρικα, έχεις το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να παρουσιάσω τις απόψεις της ε, βιομηχανίας Ντασό ε, για το θέμα το οποίο σας απασχολεί. Να υπενθυμίσω ότι το 2013 είναι μια σημαντική χρονιά γιατί υπάρχουν διάφορα ραντεβού, η επικοινωνία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Σύνοδος Κορυφής ε, του Δεκεμβρίου που θα ασχοληθεί ε, με την άμυνα στην Ευρώπη. Ως ε, Ευρωπαίος πολίτης και επικεφαλής επιχείρησης στην Ευρώπη να σας δώσω μια εικόνα της κατάστασης στον τομέα της βιομηχανίας της άμυνας και γενικά της άμυνας στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι η κατάσταση λίγο ανησυχητική. Η άμυνα, όπως ξέρετε, είναι προνόμιο των κρατών μελών και παρότι έχουμε προχωρήσει στην ΚΠΑ, ε, που δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή θέληση, η πρόσφατη εμπειρία από το Μαλί δείχνει ότι τα κράτη είναι τα υπεύθυνα για την προετοιμασία και την εξαγωγή του πολέμου. Παρότι η Ευρώπη έχει σημειώσει κάποια βήματα, κάποια πρόοδο. Επομένω, το θέμα που τίθεται είναι τι θέλουν τα κράτη στην Ευρώπη. Τι θέλουν για την Ευρώπη σε αυτόν τον ιδιαίτερο τομέα που είναι ο τομέα τη άμυνα. Ποιε είναι οι φιλοδοξίε του, μπορούμε συνέχεια να, μπορεί συνέχεια να μιλάμε για την άμυνα στην Ευρώπη, αλλά όλο και λιγότερα λεφτά δίνουμε. η κρίση είναι ένας ένοχος και για αντικειμενικούς λόγους μειώνουμε τα κονδύλια για την άμυνα. Όποιες, όποιες όμως και αν είναι οι οικονομικές συνθήκες, είτε καλές είτε κακές, εδώ και 20 χρόνια μειώνουμε τον προπολογισμό της άμυνας. Λες και οι ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι η άμυνά τους δεν είναι ευθύνη τους. Όσοι συνεισφέρουν, θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για αυτούς που συνεισφέρουν ε, και για αυτούς που κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια από άλλους. Στον τομέα της άμυνας υπάρχουν δύο δυνατότητες. Η δυνατότητα της ανεξαρτησία, ε, το να κυριαρχούμε και να ρυθμίζουμε το μέλλον μας ή ε, η απώλεια της αυτονομίας μας και της δράσης μας. Στην τελευταία περίπτωση σβήνουμε από την ιστορία, το χάρτη, φεύγει, χάνεται η κυριαρχία μας ή προσδιοριζόμαστε, προσανατολιζόμαστε σε άλλες δράσεις. Από την άλλη έχουμε την Αμερική, αύριο μεθαύριο θα έχουμε την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία ή άλλους. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ αυτό το σενάριο. Αντίθετα, ε, θέλω μια ισχυρή Ευρώπη που θα παίξει τον ιστορικό της ρόλο. Αλλά αυτή η φιλοδοξία δεν μπορεί να γίνει χωρίς τα απαραίτητα μέτρα. Γιατί η άμυνα έχει κόστος. Γιατί η κυριαρχία έχει ένα τίμημα. Εμείς δίνουμε 182 δις, ε, η Κίνα 132, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες 500 τόσα δις. Αν τα ευρωπαϊκά κράτη θέλουν να, γίνουν, να παραμείνουν εξάρτητα και να παίξουν το ρόλο τους στην ιστορία, ανάλογα με την οικονομική τους θέση, θα πρέπει οπωσδήποτε να δράσουν. Γιατί σε βιομηχανικό επίπεδο η κατάσταση που προκύπτει από αυτή την έλλειψη κονδυλίων είναι προγράμματα που έχουν όλο και λιγότερα κονδύλια, ε, απουσία νέων προγραμμάτων που δεν μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας, να διατηρήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία που είναι σε φάση οι ΙΠΑ θέλουν να εξασφαλίσουν και την οικονομική και την στρατιωτική κυριαρχία τους ε, με βάση την ε, τεχνολογική, το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, εμείς επενδύουμε πολύ λιγότερα σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Θα πρέπει στην Ευρώπη τα κράτη και η Κομισιόν όπως ακριβώς ισχύει εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, να καταλάβουν ότι η οικονομική ευημερία πάει παράλληλα με την ικανότητα προστασίας της Ευρώπης και ε, για να την εξασφαλίσουμε χρειαζόμαστε και την ανώτατη και την, την καλύτερη δυνατή τεχνολογία. Αυτό το κατάλαβαν οι ΗΠΑ και αυτό είναι σημαντικό και είναι ο καλύτερο εγγύτης για την οικονομική ευημερία, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξία της θέσης απασχόλησης και την εξασφάλιση της ηγεσία. Αυτό το κατάλαβαν, είπα, όπω είπα. Το θέμα είναι τι πολιτική αγοράς προωθούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κατάσταση των ανεπάνδρωτων εναέριων οχημάτων ε, είναι πολύ κακή για την Ευρώπη. Ε, έχει γίνει σχεδόν ταμπού αυτή η λέξη στην Ευρώπη. Είναι πολύ στρατηγικός ο ρόλος για το μοντέρνο πόλεμο με τεχνολογίες που προωθούν κυρίως στις ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν να ε, κρατήσουν το μονοπόλιο σε αυτόν τον ευαίσθητο και στρατηγικό τομέα. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος F35 που γνωρίζετε, όπου τα ευρωπαϊκά κράτη όλο ένα και πιο φτωχά θα έλεγα, έχουν δώσει μόνο 5 δισεκατομμύρια ε, δολάρια για το F-35. Ε, αυτό είναι το 80% της ανάπτυξης ε, του ποσού που χρειάζεται για ένα ραφάλι. Οι αμερικανικές επενδύσεις στα, στα drones, στα αεροπλάνα, είναι πολύ έντονες, ενώ το, εδώ στην Ευρώπη υπάρχει ένα πρόγραμμα λοιπόν στις Ηνωμένες υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την ε, επιβίωση αυτού του ε, τομέα. Στο Αφγανιστάν, στο Κόστοβο, στη Λιβύη, στο Μαλί λοιπά με διάφορες πρωτοβουλίες είδαμε πως σημαντικά, σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία. Οι προσπάθειες που κάναμε ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανία μας, επέτρεψαν να υποφεληθεί από επιπλέον πόρους. Υπάρχουν νέα διαφορετικά προγράμματα ούτω ώστε να μπορέσουν οι αμυντικές βιομηχανίες να αναπτυχθήξουν τις ικανότητές του να ενισχυθούν απέναντι στην ε, βορειοαμερικάνικη κυριαρχία και ανταγωνισμό και αύριο μεθαύριο στην παγκόσμια. Ε, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό αυτό το μέσο. Εμείς έχουμε διτές ε, δραστηριότητες και αντιμετωπίζουμε ισχυρότατο ανταγωνισμό. στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας ε, αντιμετωπίζουμε ανταγωνισμό και από τους Καναδούς και από τους Αμερικανούς. Ξέρουμε τον ανταγωνισμό. Πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Ε, έχουμε εργαλεία χάρη στα οποία κερδίσαμε αυτή τη θέση μας. Ε, μην ξεχνάτε ότι, εμείς, ε, ότι το κόστος του εργατικού, του εργατικού δυναμικού είναι πιο ακριβό εδώ. Ε, έχουμε φόρους πολύ ψηλότερους συχνά σε περισσότερες, περισσότερες χώρες από ότι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Ας μην μιλήσουμε τώρα για την Κίνα, για την Βραζιλία κτλ. Τα συγκεκριμένα μέτρα της Κομισιόν ενίσχυσαν την βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα, ερωτηματικό. Ε, το πακέτο της άμυνας με την οδηγία για τις ε, ενδοκινοτικές μεταφορές. Τι ε, επιπτώσεις υπάρχουν. Είναι σημαντικό σήμερα να αναλύσουμε αναχώρα τι συνέπειες αυτών των δύο οδηγιών. Είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά εξασφάλισαν ανταγωνιστικότητα στην, στον κλάδο. Τι θέλει τώρα η βιομηχανία. Μία αύξηση του, των κονδυλίων για την έρευνα και την τεχνολογία, την ε, εκκίνηση νέων προγραμμάτων που να βασίζονται σε αρμοδιότητες που θα μοιραστούν σε όλη την Ευρώπη. Ονειρευόμαστε η πνευματική ιδιοκτησία των ε, βιομηχάνων να γίνει σεβαστή κάτι που δεν γίνεται, δεν είναι πραγματικότητα σήμερα σε όλα τα νομοθετήματα που προωθεί η Κομισιόν ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Θέλουμε αυτή η πνευματική ιδιοκτησία να εξασφαλιστεί σε όλους τους βιομηχάνους Όταν αναπτύσσουμε μια τεχνολογία μαζί, είναι προφανέ. Αλλά όταν κάθε βιομηχανία αναπτύσσει τη δική τη τεχνολογία, αυτό δεν είναι τόσο, τόσο δεδομένο. Νομίζω ότι θα πρέπει επίση να έχουμε μια καλύτερη ισοτιμία με το δολάριο, αλλά αυτό αφορά γενικότερα την Ευρώπη. Ε, επίση, θα πρέπει να δούμε την αμοιβαιότητα, τι γίνεται σε άλλε χώρε. Δεν είναι ακριβώ η ευρωπαϊκή προτίμηση, θα πρέπει επίσης τα διάφορα αρχηγεία να βρουν κοινέ ε, επιχειρησιακές ανάγκες. Θα πρέπει να δούμε τις ε, αρμοδιότητες που έχουμε όλοι μας στην Ευρώπη για να μην φτιάχνουμε τεχνητά νέες αρμοδιότητες οι οποίες θα έρθουν σε αντίφαση και σε ανταγωνισμό με τις παλιές. Αυτά είναι από τα παράδοξα της Ευρώπης. Από τη μία δηλαδή δεν θέλουμε το μονοπόλιο, από την άλλη Μιλάμε για την ενίσχυση του αμυντικ... της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτά τα θέματα θέλουμε να τα συζητήσουμε λοιπόν. Για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Τι μπορούμε να ζητήσουμε εμείς οι, βιομηχανοί. Καταρχάς, πρώτο σημείο, όχι νέε οδηγίες. Νομίζω ότι πρέπει να αναλύσουμε τις ισχύουσες. Δεν είναι το νομοθετικό πλαίσιο που θα χτίσει την Ευρώπη της της Επίσης, η ασφάλεια του ανεφοδιασμού είναι καλό πράγμα, θα πρέπει να το προωθήσουμε, αλλά όπως ακριβώς το κάνουν και οι Αμερικάνοι για τα δικά τους προϊόντα. Τρίτον, ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα, νομίζω ότι πρέπει πάνω απ' όλα να ενισχύσουμε τη ζήτηση και την, ε, την ε, εναρμόνιση των ευρωπαϊκών αναγκών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ο Οργανισμός Άμυνας θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το ρόλο. Να ενισχύσουμε, να εντοπίσουμε τα κέντρα αριστείας και εδώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας θα μπορούσε να δώσει συμβούλια, να κάνει μια χαρτογράφηση, να δει πού υπάρχουν πραγματικά οι αρμοδιότητες αυτές, να βασιστούμε σε αυτές και εκεί να ρίξουμε χρήματα, όπου υπάρχουν ήδη ε, προσόντα αρμοδιότητες. Φυσικά να δώσουμε λεφτά στην ε, έρευνα και στην τεχνολογία. να μπει και ο τομέας της άμυνας ε, στα διάφορα προγράμματα με τους κανόνες που πρέπει, όπου οι επενδύσεις των επιχειρήσεων θα καταλαβαίνετε ότι, πρέπει ότι δεν μπορεί να είναι άπειρες, γιατί πρέπει μετά να αποδώσουν ε, αυτές οι επενδύσεις. Αυτές είναι κάποιες από τις προτάσεις του κλάδου. Το τελευταίο σημείο είναι ότι μας ανησυχεί λιγάκι η θέληση. Του να μπει, η θέληση που υπάρχει στην Ευρώπη να μπει το θέμα της άμυνας στο Free Trade Agreement. Για να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να είμαστε ισότιμοι. Θα πρέπει καταρχάς πρώτα να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία πριν μιλήσουμε ισότιμα με την αμερικανική βιομηχανία, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύουμε να μας φάνε λάχανο. και να γίνουμε απλοί υπεργολάβοι. Κι όμως η Ευρώπη με το κόστη που έχει αποκλείεται να επιβιώσει ως υπεργολάβος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθήσουμε τις δικές μας τεχνολογίες. Ένα μικρό συμπέρασμα τώρα. Νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να, προωθήσουμε και να λανσάρουμε νέα προγράμματα. Η Κομισιόν μπορεί να βοηθήσει εδώ. Μπορεί να δώσει ε, τα λεφτά στην έρευνα και στην τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα μπορεί να βρει τι καλέ περιοχέ, του καλού βιομήχανου που θα κάνει. Θα παίξει το ρόλο του. Ο καθένα θα παίξει το ρόλο του. Αλλά βεβαίω πάνω απ' όλα είναι τα κράτη. Τα κράτη έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν νέα προγράμματα, να δρομολογήσουν νέα προγράμματα. Και όπως αυτό που έγινε στη συνθήκη του Λάγκεστερ, Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δύο χώρες που είναι πρωτοπόροι. Αν θέλουν να έρθουν και να συνταχθούν με εμάς, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, ε, οι χώρες του Βορρά, ε, είναι χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Γαλλία. Αλλά χρειάζεται μια ατμομηχανή. Λεφτά. Ετοιμάζω τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις αναπτύσσω τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μπορώ να μπω πρώτος σε μια σύραξη, ε, συνεισφέρω, ο καθένας όσο μπορεί, με πραγματικά, πραγματικά συνεισφέρω, με τα απαραίτητα ποσά και η λύση είναι να είμαστε ε, ρεαλιστές και να λειτουργούν όλα αυτά με μεταβλητή γεωμετρία, όπως ακριβώς πρέπει. Σας ευχαριστώ. Έχω αρκετές ερωτήσεις να θέσω. Θα το δούμε αργότερα αυτό και στις ε, ερωταπαντήσει με τους συναδέλφου. Από την Αγκούστα Γουέστλαν, τον κύριο Ρωμητή. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε ε, να μιλήσω και να ακούσετε κι εσείς τον κλάδο. Όπως είπε ο κύριος Τχαπιέ, όπως είναι και καταφανές, ζούμε σήμερα σε μια πολύ διαφορετική Ευρώπη από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Η οικονομική κρίση του 2008 ε, άλλαξε τελείως τα δεδομένα στην ε, παλιά ήπειρό μας. Και οι ευρωπαϊκές χώρες ε, δυσκολεύονται όλο και πιο πολύ να αναπτύξουν ένα αυτόνομο, ένα στρατιωτικό πρόγραμμα. κάτι, αυτό κάτι ήταν, ε, παλιότερα ήταν κάτι πολύ πιο νεφελώδες, ναι, αλλά σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Και αν θέλουμε η ευρωπαϊκή βιομηχανία όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να ανταγωνιστεί με τους, διε, τους διεθνείς εταίρους, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Γιατί αν συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε μόνο σε εθνικό επίπεδο, με όλα τα όρια που συνεπιφέρει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε προτάσεις και να φτιάξουμε ε, πραγματικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν μειώσουμε τα κονδύλια στην έρευνα και στην ανάπτυξη στην Ευρώπη, τότε θα στείλουμε την αμυντική βιομηχανία σε μια σταθερή και αδυσόπιτη ύφεση από την οποία θα μπορεί να εξέλθει. Τα προγράμματα, τα, η τεχνογνωσία μας βασίζονται σε σημαντικές επενδύσεις που κάναμε τα περασμένα χρόνια στην έρευνα και στην τεχνολογία. Ε, τα τελευταία 20 χρόνια. Κάναμε τρομερές προσπάθειες. Αν δεν συνεχίσουμε θα χάσουμε εντελώς την αυτονομία της αμυντικής μας βιομηχανίας. Είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμήσουμε αυτή την τάση όταν δεν έχουμε αντίστοιχα εργαλεία όπως οι ΗΠΑ, όπου ε, το πρόγραμμα για, το, για τα rotorcraft είναι βασικό κλειδί για τη μελλοντική ανάπτυξη. Εμείς βλέπουμε τις ε, ο, όλο και πιο επιθετικές πολιτικές των Αμερικανών στην, στον τομέα της αεροναυπηγικής. Έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Το Foreign Military Sales, παραδείγματο χάρη, ένα πολύ σημαντικό. Με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι τώρα αρχίζει να αντιδρά κάπως η Ευρώπη. Ε, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια, ε, θα υπάρξει και η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφή το Δεκέμβριο που θα ασχοληθεί με την Ευρωπαϊκή Άμυνα με το σκοπό να βελτιώσουμε τις στρατιωτικές ε, δυνατότητες της Ευρώπης και να ενισχύσουμε την ε, αμυντική μας βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας προωθεί διάφορες πρωτοβουλίες. Έχουν την Task Force που προωθούν οι αρμόδιοι επίτροποι. Είναι θετικές αυτές οι πρωτοβουλίες. Όπως και το pooling και sharing ε, που όμω υπολείπεται πάρα πολύ σε σχέση με αυτά που πρέπει να κάνουμε και να τα κάνουμε γρήγορα. Συνάδελφοι και αγαπητοί ευρωβουλευτές, εγώ είμαι Γενικός Διευθυντής τη Αγκούστα Westland και νομίζω ότι στον τομέα των ελικόπτερων ε, έχουμε πραγματικά το κλειδί της αριστείας. Ε, θα σας μιλήσω για τον τομέα του Rotocraft Industry, όπου παίζουμε καθημερινά εμείς. Είμαστε ηγέτες στον εμπορικό τομέα, στην εμπορική αγορά, που είναι ανταγωνιστική και ανοιχτή, εξορισμού. Αν λάβουμε υπόψη μας τη διάσταση της αγοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί έχουμε μια καλή θέση. Αλλά ακόμα και σε σχέση με αυτό έχουμε καλή θέση και σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι η Αγκούστα Westland είναι στον τομέα των, αυτών των ελικόπτερων, το Rotocraft, έχουμε ηγετικό ρόλο. Έχουμε μία σειρά από στρατιωτικά και εμπορικά ελικόπτερα και δεν υπολοιπόμαστε σε καμία περίπτωση ε, σε σχέση με τους Αμερικανούς και σε αυτό που μπορούν να προσφέρουν. Η Αγκούστα και η Westland μαζί έχουν αναπτύξει ε, το ελικόπτερο των 11 τόνων, που είναι ένα ελικόπτερο από τα πιο εξελιγμένα τα τελευταία χρόνια. Και επενδύουμε για να προσαρμόσουμε την τεχνολογική μας πραγματικότητα στην εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς. Σε ορισμένε περιπτώσεις η Αγούστα η Augusta Westland ε, προλαβαίνει τις νέες ανάγκες και συχνά και συνέχεια επενδύουμε ένα πολύ σημαντικό τμήμα των εσόδων μας. Ε, το 12% ε, πηγαίνουν στην, ε, είναι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Για να σας πω, τα τελευταία λιγα λίγα χρόνια, 4-5 χρόνια ας πούμε, επενδύσαμε σε πάνω από 6 καινούργια μοντέλα. Το 159, ένα άλλο που φτιάξαμε μαζί με την τουρκική βιομηχανία, το 149 που είναι ένα μοντέλο στρατιωτικό στην ε, κατηγορία Utility Transport και έχουμε εισαγάγει και άλλα τρία μοντέλα, το 139 στις 6,5 τόνους, το 169 και άλλο ένα. Για να σας δείξω ότι δεσμευόμαστε και θέλουμε πραγματικά να παραμείνουμε ηγέτες ε, στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτά τα ελικόπτερα, αυτή η τελευταία γενιά ελικόπτερων, για πρώτη φορά εισάγει στην βιομηχανία μας μια νέα αντίληψη της ε, τεχνολογικής οικογένειας, ε, μια νέα έννοια. Δηλαδή, θέλουμε να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, να περνάνε από το ένα μοντέλο στο άλλο. Και αυτή την έννοια της ε, οικογένειας την εφαρμόζουμε, της εμπορικής οικογένειας ας πούμε, την εφαρμόζουμε και στα στρατιωτικά ελικόπτερα λαμβάνουμε υπόψη μας την οικονομική κατάσταση των στρατών μας, των ενόπλων δυνάμεών μας. Και θέλουμε, λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την κατάσταση, να τους δώσουμε το καλύτερο δυνατόν προϊόν. Ε, προϊόντα, η ίδια οικογένεια έχει την ίδια φιλοσοφία, τα ίδια συστήματα, την ίδια υποστήριξη και, την, και το training βέβαια. υπάρχει μια συζήτηση ε, για τη χρήση της λεγόμενης διτής τεχνολογίας. Δηλαδή μια τεχνολογία που μπορεί να εφαρμοστεί και στον εμπορικό τομέα και στο στατιωτικό τομέα. Και εμείς, ε, η εταιρεία μας δηλαδή, ε, πιέζουμε, προωθούμε, ούτως ώστε αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε εδώ και λίγα χρόνια να προχωρήσει και να προλάβει την εξέλιξη της αγοράς. Επίσης, μια και είναι λίγα τα κονδύλια, θα πρέπει να ξοδεύονται με σοφροσύνη. Αυτή η έννοια της ε, οικογένειας, ακριβώς, λαμβάνει υπόψη την ε, σπάντα των πόρων. Αυτή η έννοια της δυτής τεχνολογίας μπορεί να εφαρμόσει, μπορεί να μας εξασφαλίσει και οικονομίες κλίμακας επίσης. Η Αγκούστα επίσης προβλέπει τις εξελίξεις των ε, μελλοντικών ελικόπτερων. Ε, αναπτύσσουμε το ε, ελικόπτερο 609. Ε, στην αρχή ε, είχαμε ένα joint venture με τους Αμερικάνους και εν συνεχεία αγοράσαμε το πρόγραμμα από εκείνους. Το 609, το ελικόπτερο 609 είναι ένα ελικόπτερο, ένα αεροπλάνο που μπορεί να απογειωθεί και να προσγειωθεί κάθετα και μπορεί να πετάξει σε πολύ μεγάλο ύψος έχει... και μπορεί να πετάξει στο διπλάσιο της ταχύτητας και του βελινεκούς αν το συγκρίνουμε με τα κλασικά ελικόπτερα. Εμείς λοιπόν πιέζουμε να μπει αυτό το μοντέλο σε παραγωγή και ταυτόχρονα διερευνούμε νέες ε, εφαρμογές πιο προηγμένες που βασίζονται πάντα σε αυτή την τεχνολογία του Tilt Rotocraft. Και... και μπορούν να κάνουν πράγματα που κάνουν αεροπλάνα 20 θέσεων. Έχουμε το πρόγραμμα Clean Sky προωθώντας αυτή την τεχνολογία για να προωθήσουμε αυτή την μορφή ελικόπτερων. Είναι πολύ, είμαστε πολύ δραστήρια. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν πολλά, πολλή ζήτηση για το Rotocraft και ε, από τις ναυτικές δυνάμεις και από τις χερσαίες δυνάμεις. Να τονίσω και κάτι άλλο για την Augusta Westland. Συχνά συζητάμε το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το βιομηχανικό τομέα, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το πλεονάζον δυναμικό και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Η Αγκούστα Westland προώθησε ε, μια πολύ ένα πολύ σημαντικό, μια... ένα παράδειγμα θέλετε, διεθνοποίησης. Κάναμε μία κοινοπραξία ανάμεσα σε μία Ιταλική εταιρεία την Αγκούστα και μία Αγγλική την Westland. Τον 20ο αιώνα ενισχύσαμε αυτή την συνεργασία ε, προσθέτοντας ε, στην κοινοπραξία αυτή και την πολωνική εταιρεία ελικοπτέρων. Έχουμε τρεις χώρες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται και μάλιστα ε, μια αμερικανική μονάδα στη Φιλαδέλφια που ανήκει στην εταιρεία μας παράγει τα εμπορικά ελικόπτερα. Επομένως προλάβαμε τις ανάγκες των κυβερνήσεων ό,τι αφορά την ενοποίηση. Και η γυροκόπια είναι παράδειγμα αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, Εκεί έχουμε συνεργασία ε, Γάλλων και Γερμανών. Ε, συνεχεία προσθέθηκαν και οι Ισπανοί. Οι Ισπανικές εταιρείες ελικόπτερων. Τι χρειαζόμαστε. Η Ευρώπη θα πρέπει πιο εντατικά και καλύτερα να υποστηρίξει αυτές τις τεχνολογίες αεροναυπηγικής και διαστήματος που σήμερα ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα για ελικόπτερα στρατιωτικά που να δρομολογείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο με το GMR των Ηνωμένων Πολιτειών που δρομολόγησαν πολύ πρόσφατα. Εμείς θα πρέπει λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μας, να κάνουμε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια. Θα πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινότητα που θα πρέπει να ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα και να καλύψει αυτό το τεράστιο κενό που υπάρχει σε σχέση με τους Αμερικάνους. Αν αναπτύξουμε αυτή την τεχνολογία διτής χρήσης, το Dual Use Technology, με έξυπνες δαπάνες, μπορούμε να αναπτύξουμε με ανταγωνιστικό τρόπο τη βιομηχανία μας, ούτως ώστε αυτή η τεχνολογία, η ίδια τεχνολογία, να μας επιτρέψει να ανταγωνιστούμε στην παγκόσμια αγορά. Φυσικά υπάρχει και μια αναδυόμενη ανάγκη εξορθολογισμού ε, και ενσωμάτωσης των προγραμμάτων ε, προμήθειας, καθώς και του σχεδιασμού των προμηθειών. Ευχόμαστε σε αυτό το τομέα να παίξει όλο και πιο φιλόδοξο ρόλο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο ετήσιος προπολογισμό της είναι 30 εκατομμύρια μόνο. Επομένως δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχει τη δυνατότητα να προωθήσει αυτά τα μεγάλα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, ε, κάναμε μια προσπάθεια εξορθολογισμού της ε, πολιτικής μας και της παραγωγής μας και η Αγκούστα Westland με την συγχώνευση σημαντικών ευρωπαϊκών ε, βιομηχανιών ελικοπτέρων έκανε την προσπάθειά τη. Ο καθένα θα πρέπει να λάβει τι ευθύνε του. Ε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για ευρωπαϊκή άμυνα αν προβλέπουμε συνέχεια περικοπέ στην έρευνα και την ανάπτυξη. Πώ μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αν υπάρχουν χώρε ε, που σε εθνικό επίπεδο δεν ε, συνεργάζονται. Η έρευνα και η ανάπτυξη όχι μόνο πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά θα πρέπει βεβαίω να ξοδεύουμε καλύτερα, πιο έξυπνα και εδώ είναι μια άλλη συζήτηση όμω και δεν νομίζω ότι είναι το κατάλληλο βήμα. Χρειαζόμαστε όμως τα ευρωπαϊκά όργανα να μας διευκολύνουν σε ό,τι αφορά τον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας κάνω μία σύσταση. Στην Ευρώπη σίγουρα υπάρχει ανάγκη ε, πιο προσεκτικού, ε, προσεκτικής ρύθμισης σε ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα, με εστίαση ειδικά στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να δούμε πώς γίνονται οι κανόνες, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα προγράμματά μας, ε, δίνοντας τη δέουσα προσοχή και στην πνευματική ιδιοκτησία, στα πνευματικά δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εγώ υποστηρίζω την ευρωπαϊκή βιομηχανία και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί μας διαφωτίσατε και εσείς ε, ε, για το θέμα αυτό και υπήρχαν και κάποιες ε, διαφορές ε, σε, σχέση με τον πρώτο καλεσμένο μας, ε, ιδιαίτερα για τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στα θέματα αυτά θα επανέλθουμε και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάνν Πίε, just starting this... προσπαθώ να ξεκινήσω με τις διαφάνειες. Για να δούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου παράλληλα με τις διαφάνειες, αν γίνεται. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, παρακαλώ. Can you, can you just make it... F5. F5. F5. Okay. Yeah, okay. So, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που λαμβάνω το λόγο εδώ εκ μέρους της Σουηδικής Ένωσης Βιομηχανιών Ασφάλειας και Άμυνας, γιατί πραγματικά έχουμε τεράστιες προκλήσεις στην Ευρώπη, αλλά και για την βιομηχανική βάση μας για την ασφάλεια και άμυνα αυτές τις μέρες ε, των εύλογων ανησυχιών και τις κατήφιες και τους ζώφους θα κάνω την μπορώ για να δώσω μια θετική νότα για τις προοπτικές, ε, το μέλλον και τις δυνατότητες που έχει η ευρωπαϊκή αυτή βάση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, παρουσιάσω τις εμπειρίες μου από τη ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα στην Σουηδία για την ε, βιομηχανική βάση της ασφάλειας και άμυνας. Έτσι τροποποιήθηκε η προσέγγισή μας και άλλαξε και γνώμη στο πώς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσεγγίσει αυτό το θέμα. Θα σας ε, κάνω μια παρουσίαση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο τομέα αυτό και τέλος θα σας κάνω κάποιες προτάσεις ε, για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με αποτελεσματικό τρόπο. Όλα αυτά με πρόθεση να έχουμε μια επιτυχή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση για την ασφάλεια και την άμυνα κατά τον 21ο αιώνα. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Άμυνας είναι ένα θέμα κεφαλαιόδου σημασίας, όχι μόνο για όσους εργαζόμαστε στον κλάδο αυτό, αλλά για το σύνολο του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τοπίου. Και θα τολμούσα να πω ακόμη και για το μέλλον μιας ανταγωνιστικής, ασφαλούς και ευημερούσας Ευρώπης. Η Σουηδία ε, ξεχωρίζει κατά κάποιο τρόπο στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό τοπίο άμυνας, ε, τουλάχιστον για τρεις λόγους. Πρώτον, η Σουηδική βιομηχανική βάση είναι σχετικά και μεγάλη και επιτυχής, αλλά και στραμμένη προς τις εξαγωγές. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο με συγκρίσιμο μέγεθο και οικονομία δεν μπορεί να δώσει τέτοιε πλατφόρμες συστήματο στον αέρα, ξηρά και θάλασσα. Είναι μία από τι 7 χώρε στον κόσμο που κατασκευάζει πολεμικά αεροσκάφη. Και μια και η βιομηχανία αυτή εργαζόταν με ένα σχετικά μικρό πελάτη, όπω ήταν οι Σουηδικέ Ένοπλε Δυνάμει, η σχέση κόστου-οφέλου ήταν πολύ σημαντική για όλε τι τεχνικέ λύσει. Κάτι που μα έκαναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικού ε, και ιδιαίτερα τώρα σε εποχέ λιτότητα. Η Σουηδία, με βάση το Ινστιτούτο τη Στοκχόλμη για την έρευνα στην ειρήνη, είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέ αμυντικού εξοπλισμού κατά κεφαλήν στον κόσμο το 2011 και μάλιστα οι εξαγωγέ αυξήθηκαν κατά 400% την τελευταία δεκαετία. Βέβαια, η εγχώρια αγορά ε, ε, θεωρείται ως μία ακόμη αγορά από τις Σουηδικές εταιρείε. παρόλο που είναι πολύ σημαντική αυτή η εγχώρια αγορά, γιατί ε, είναι σημαντική και ως σημείο αναφοράς. Ε, επίσης, γινόμαστε όλο και λιγότερο εξαρτημένοι από την ευρωπαϊκή αγορά και προσανατολισόμαστε περισσότερο στις αναδυόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα της Ασίας. Έτσι συνδυάζουμε τις εξαγωγές μας με ένα πολύ αυστηρό, από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου των εξαγωγών στον κόσμο. Δεν θεωρούμε ότι αυτό το αυστηρό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών είναι ένα άχθος. Αντίθετα, είναι ένα πλεονέκτημα, ένα ατού για τη βιομηχανία, γιατί παρέχει νομιμοποίηση και αποτελεί προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε μεταφορές τεχνολογίας, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένε Πολιτείες, που είναι απαραίτητος εταίρος για τη Σουηδία παρά τι τεράστιε προκλήσει που δημιουργεί η νομοθεσία ΙΤΑΡ, θα ήθελα να πω εμπαρόδο. Κατά τη γνώμη μου, η επιτυχία στι διεθνείς αγορέ και μια φιλόδοξη προσέγγιση στον έλεγχο των εξαγωγών είναι, κάτι, είναι θέματα αλληλένδετα μεταξύ τους και άρρηκτα συνδεδεμένα. Δεύτερον, η Σουηδική Βιομηχανική Βάση Ασφάλεια και Αμυνα είναι η μοναδική στην Ευρώπη, μεγάλη σημασία, που ε, ανήκει αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι και αλλοδαπή ιδιοκτησία. Αυτά μια στρατηγική απόφαση που έλαβε το Σουηδικό Κοινοβούλιο στη δεκαετία του 90 και μάλιστα η βιομηχανία εκτιμά ιδιαίτερα αυτή την επιλογή. Για να το πω απλά, οι κυβερνήσει ε, δεν διαχειρίζονται καλύτερα τι ε, βιομηχανίε Άμυνα από ότι οι ιδιώτε. Επιπλέον, το γεγονό ότι έχουμε και άλλο αλλοδαπή κυριότητα μα κάνει πιο προσάρμοστου ε, στι εκστρατείε χρηματοδότηση και πωλήσεων σε δύσκολου καιρού. Έχουμε μεγαλύτερε συνεργασίε σε διεθνή σχέδια και καλύτερη πρόσβαση στι διεθνεί αγορέ. Σε καμία περίπτωση αυτή η ιδιωτική ιδιοκτησία δεν οδηγεί σε μετακατάσταση ε, των επιχειρήσεων από τη Σουηδία. Το αντίθετο, ο αριθμό των απασχολούμενων στη Σουηδική βιομηχανία άμυνα ε, βρίσκεται σχεδόν στο απόγειο τη σήμερα. Και μάλιστα μέσα σε μία δεκαετία ε, έχουμε μείωση κατά 15% των της, ε, των δημοσίων προμηθειών υλικού, ενώ της, α, ε, ε, των σουηδικών πωλήσεων το ποσοστό αυξήθηκε κατά 44%. Είμαστε επίσης, επαιδείουμε ιδιαίτερη στην στην ε, έρευνα. Η ΣΑΜΠ, ο μεγαλύτερος όμιλος, ε, ε, επενδύει το 25% του τζίρου της σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και 18% του 3,5 δισεκατομμύριο του τζίρων των σουηδικών εταιριών επενδύεται σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτό, σε αυτό μας βοηθά βέβαια και η ακμαία επιστήμη και τεχνολογική, επιστημονική και τεχνολογική μας βάση. Μάλιστα, ο δείκτης του ΩΣΑ δείχνει ότι έχουμε τα περισσότερα ε, διδακτορικά σε επιστημονικά και τεχνολογικά σχέδια. Έχουμε επίσης ε, Είμαστε τρίτοι στον ΩΣΑ σε ό,τι αφορά την ποιότητα των τεχνολογικών, τεχνικών μας, πανεπιστημίων και σχολών. Τώρα, να μιλήσω και λίγο για τι προκλήσει τη Ευρώπη. Κανένα νησί δεν είναι απομονωμένο. Κανένα έθνο δεν είναι νησί. Κανένα έθνο δεν είναι απομονωμένο σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και παρά την ροδαλή εικόνα που σας έχω δώσει για την ε, σουηδική βιομηχανία, σίγουρα και εμείς επηρεαζόμαστε και ανησυχούμε τα μάλλα για την οικονομική ύφεση της Ευρώπης. Βέβαια, Ομολογούμε ότι οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση ασφάλειας και άμυνας είναι πολύ παλιότερες από το 2008, την στιγμή της κρίσης δηλαδή. Γιατί για δεκαετίες είχαμε κατάσταση υπερπαραγωγής. δεν είχαμε οικονομίες κλίμακος και επίσης είχαμε και περιττή επικάλυψη σε ό,τι αφορά τον αμυντικό αξιοπλισμό ενώ δεν έχουμε βασικές τεχνολογίες διαχείρισης στρατιωτικής διαχείρισης των κρίσεων, κάτι που μας δημιουργεί προβλήματα στην παρουσία μας ε, ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και η εμπειρία μας από τη Λιβύη και το Μάλι είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της αδυναμίας. Επίση, λόγω τη κρίση και τη οικονομική ύφαση, είχαμε δραστική περικοπή των αμυντικών δαπανών, κάτι που δημιουργεί μια ανυπόφερη κατάσταση. Αν δεν μεταρρυθμίσουμε τι δημόσιε προμήθειε και δεν ανοιχτούμε στον ανταγωνισμό στην Ευρώπη, θα χάσουμε τι δυνατότητέ μα, όχι εξαιτία τη συρρήκλωση μόνο των αμυντικών μα προπολογισμών, αλλά και εξαιτία ότι αποδεχόμαστε πολύ δυσμενεί σχέσει κόστου-οφέλου οι βιομηχανίε θα υποφέρουν αν χάσουμε τέτοιε δυνατότητε. δυνατότητες. Ακόμη και οι πιο ανταγωνιστικές εταιρείε θα πρέπει να περιοριστούν. Θα πρέπει να ε, επαναπροσανατολιστούν σε άλλους τομείς, κάτι που μπορεί να έχει ε, δυσμενείς επιπτώσεις στον τομέα τη άμυνας. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν μπορούν πια να ξοδεύουν χρήματα που δεν έχουν για πράγματα που δεν χρειάζονται μάλιστα, που τους είναι περί τα εξαιτίας του προστατευτισμού. Σέβομαι την άποψη εκείνων που λένε ότι η διαχείριση μιας διαδικασίας μεταρρύθμισης ε, στο βιομηχανικό αμυντικό τομείο και άνοιγμα στο περισσότερο, σε περισσότερο ανταγωνισμό ε, θα δημιουργήσει τον κίνδυνο ανεργίας ιδιαίτερα στην εποχή της λιτότητας και της ύφεσης. Δεν συμφωνώ όμως με τη γνώμη αυτή, παρόλο που τη σέβομαι. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που περισσότερο χρειαζόμαστε στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή η ανταγωνιστικότητα και μια βιώσιμη ευημερία. Ε, θα θυμάστε ότι την ελληνική την ευημερούσα Ευρώπη την οικοδομήσαμε κατεδαφίζοντας τείχους, έρωτας δασμολογικούς και εμπορικούς φραγμούς και με ένα άνοιγμα προς τον ανταγωνισμό τέτοιες περιστάσεις χρειαζόμαστε και στην αγορά της άμυνας, γιατί εκεί οι πελάτες μας είναι μόνο τα κράτη. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε και το θέμα της ασφάλειας των εφοδιασμού και το ζήτημα της αυτονομίας. Οι βασικοί παράμετροι όμως της οικονομίας της αγοράς λειτουργούν και στον αμυντικό τομέα. Και νομίζω ότι θα ξεγελούσαμε τον εαυτό μας αν ισχυριζόμασταν κάτι διαφορετικό. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για το ποιο είναι ο ακολουθητέο δρόμο, η ακολουθητέα πορεία και τι κατά τη γνώμη θα πρέπει να κάνουμε. Τέσσερα είναι τα βασικά μου σχόλια και προτάσει. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τι ικανότητε και του συντελεστέ, του διάφορου παράγοντε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει την ανακοίνωσή τη ε, εν ώψη τη Συνόδου Κορυφή ε, των Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων που θα λάβει η χώρα το Δεκέμβριο. Και μάλιστα μερικοί φοβούνται ότι ε, θα είναι αρνητική μια υπερβολική εισχώρηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα χωράφια τη ασφάλεια και τη άμυνα και ιδιαίτερα στο θέμα του εμπορίου. Εγώ δεν συμφωνώ. Α είμαστε ειλικρινεί. Οι προηγούμενε προσπάθειε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει τη υπερπαραγωγή, τη έλλειψη οικονομία κλίμακο και του προστατευτισμού έχουν αποτύχει. Ούτε τα κρατη Ούτε η κοινή δήλωση προθέσεων των έξι εθνών, ούτε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, ούτε η Ένωση Αεροναυπηγική Διαστήματος και Άμυνας κατάφερε να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο ε, βιομηχανικό επίπεδο άμυνας ή ένα πεδίο ίσων και θε, και θεμητού ανταγωνισμού. Αν τα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα την υποστηρίξω ολόθερμα. Δεύτερον, βασικές νομοθετικές διατάξεις της αγοράς ήδη υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό και ε, στην Ευρώπη με το πακέτο της άμυνας. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερη νομοθεσία, αλλά πιο αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουμε εφαρμογή, σωστή εφαρμογή της ε, νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, προκειμένου να επιτύχουμε στο έπακρο οικονομίας κλίμακος στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε μια εναρμόνιση των κριτηρίων και εδραίωση της ζήτησης σε όλους τους τομείς στρατηγικής σημασίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν με σαφήνεια τις ε, βασικές τους ε, δυνατότητες άμυνας που θα πρέπει να υποστηριχθούν από μια ε, ρωμαλαία και οικονομική στρατηγική ασφαλεία ε, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, Φυσικά με βάση του ειδικού κανόνε εσωτερικής αγορά που ισχύουν για την άμυνα, κάτι που θα εξασφαλίσει συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ε, ανάπτυξη και διατήρηση τεχνολογιών εχμής και ιδιαίτερες ερευνητικές προσπάθειες και προσπάθειες τεχνολογικής ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα χρήματά μας ώστε να πιάσουν τόπο αποφεύγοντας ε, τον κατακαιρματισμό ε, των ερευνητικών προγραμμάτων και κάνοντας μια καλύτερη εράρξη των προτεραιοτήτων μας. Και μάλιστα το ισχύον σύστημα για τον ε, ορίζοντα 2020 είναι υπερβολικά περίπλοκο και επαχθές. Θα επιβραδύνει και δεν θα βοηθήσει καμία περίπτωση την αμυντική βιομηχανία. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά την ε, εγκαθίδρυση κέντρων, εξοχή, ε, ε, κέντρων αριστείας ή στρατηγικών πόλων, θα πρέπει να μην δημιουργούνται από πολιτικές μόνο προθέσεις και σχεδιασμούς, αλλά να προσανατολίζονται προς την αγορά. Μόνο έτσι θα είναι ανταγωνιστικά τα κέντρα αυτά αριστείας και βιώσιμα. Και μάλιστα, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τα χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Συνοχής, για παράδειγμα, θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Καταλήγοντας λοιπόν σε κάποια συμπεράσματα, ε, θα ήθελα να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Ε, το όραμά μου για περισσότερο ανταγωνισμό και συνθήκε ισότητα ανταγωνισμού στην Ευρώπη θα είναι αρκετά επώδυνο και θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι στη βιομηχανία. Αλλά αν δεν ανταπεξέλθουμε στι υφιστάμενε προκλήσει, η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Γιατί είχαμε συνηθίσει σε μια ιδιαίτερα ισχυρή ευρωατλαντική κυριαρχία στον τομέα αυτό. Με τι ευρωπαϊκέ και αμερικανικέ εταιρείε να ε, αντιπροσωπεύουν το 80% του συνολικού τζίρου της αμυντικής βιομηχανίας. Τώρα θα πρέπει να ετοιμαστούμε για κάτι καινούργιο, γιατί νέες βιομηχανίες αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς από αναδυόμενες οικονομίες, καθιστώντας πολύ πιο έντονο τον ανταγωνισμό για το μέλλον. Αν λοιπόν μπούμε σε αυτό το καινούργιο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς προηγουμένως να έχουμε ολοκληρώσει την απαραίτητη αναδιάρθρωση στην Ευρώπη, θα βγούμε όλοι χαμένοι στο τέλος. Ίσως δημιουργηθεί ένα σενάριο ε, πολύ ζωφερό με απώλεια θέσεων και διαφυγή τη έρευνα και τη τεχνολογική ανάπτυξη εκτό Ευρώπη. Αν αντίθετα ανταπεξέλθουμε στι προκλήσει, κάνουμε ένα άνοιγμα προ τον υγιή ανταγωνισμό, ξοδέψουμε χρήματα με πιο ιεραρχημένο τρόπο και σε στρατηγικά σχέδια που θα δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικές και αποδοτικέ στρατηγικές ικανότητε και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τότε έχουμε κάθε ευκαιρία για επιτυχημένη ασφάλεια και επιτυχή ε, βιομηχανική αμυντική βάση και στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Βλέπω ότι πολλοί ευρωβουλευτές ζήτησαν το λόγο μετά από τον πρώτο γύρο των ομιλιών. Θα ακούσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μέλινγκ για τη δική του παρουσίαση. Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις. Η μία π.χ. τις προηγούμενες μας συζητήσεις, τις συζητήσεις προηγούμενης εβδομάδας με θέμα τις ευρωατλαντικές σχέσεις και το ευρωατλαντικό εμπόριο σε θέματα άμυνας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τη δική σας γνώμη γιατί και για το και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γεγονό ότι συμπεριλαμβάνεται και η άμυνα στην διαπραγματευτική εντολή θα επιτρέψει στι αμυντικέ βιομηχανίε Ευρώπη να έχουν καλύτερη πρόσβαση στι αμερικανικέ αγορέ. Πολύ καλύτερη από ό,τι σήμερα. Πολλοί μίλησαν ε, για ανεφοδιαστικά αεροσκάφη και έδωσαν και άλλα παραδείγματα ε, όπως στο παρελθόν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ε, ε, προσέκρουσαν σε εμπόδια και με μια συμφωνία ελεύθερων ε, συναλλαγών ίσως τα εμπόδια αυτά αρθούν. Είστε κι εσείς αυτής της γνώμης ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Για τα ντρόν, τα μη επαδρομένα αεροσκάφη. Συζητήσεις γίνονται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για προγράμματα που ξεκίνησαν αλλά δεν ευωδόθηκαν, για άλλα προγράμματα που δεν ξεκίνησαν καν για την αγορά από τη Γαλλία αμερικανικών τέτοιων μη επαδρομένων αεροσκαφών, drones. Θα ήθελα λοιπόν να, ρωτήσω τον πρόεδρο αυτής της πολύ γνωστής αεροναυπηγικής εταιρείας ε, τη γνώμη του. Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό βραχυπρόθεσμα και ένα μεσοπρόθεσμα ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την κατασκευή τέτοιων μη επαδρομένων αεροσκαφών. Πιστεύετε ότι τέτοιες πολιτικές αποφάσεις ε, μπορεί να ληφθούν ακόμη και από τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Αυτές είναι οι δικές μου ερωτήσεις και τώρα θα δώσω το λόγο στον Μίχαλ Γκάλερ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση από τις διαφορετικές χώρες, αλλά εκάστοτε από πλευράς της ε, αρμόδιας βιομηχανίας ή βιομηχανικών κύκλων και με αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας από το Ευρωκοινοβούλιο για τη σύνταξη για αυτό το θέμα από πλευράς μας, έχω φυσικά εδώ τη διεκδίκηση, την απέτηση να βρούμε μια ευρωπαϊκή πρόπτικη που θα παρουσιάσουμε. Και συνειδητοποιώ πάρα πολύ καλά φυσικά το ότι η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια που στις επιμέρους χώρες ενδιαφέρθηκαν για τις επιμέρους βιομηχανίες, εθνικές βιομηχανίες, πολιτικοί που ήθελαν να επανεκλέγονται ή στις δικές τους περιφέρειες είχαν κάποιες βιομηχανίες. Αυτή ήταν η επιθυμία και ο στόχος τους κυρίως, να μεριμνούν ώστε τίποτα να μην αλλάξει και να μην συμβεί κάτι και πάει στραβά. Και σίγουρα επί πολλά χρόνια αυτό συνεχίστηκε έτσι με πολύ εθνικό χαρακτήρα από πλευράς προσέγγισης και επί πολλά χρόνια μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό γιατί υπήρχαν αρκετά χρήματα για να γίνει αυτό και έτσι αγνοούσαμε τους άλλους ή τουλάχιστον δεν επιθυμούσαμε να είχαμε κάποια ανεπιθύμητη ανταγωνιστική τάση που θα δυσχαίραινε τη ζωή μας. Υπάρχει και μια άλλη κατάσταση σήμερα και συνολικά μια διαφορετική κατάσταση όσον αφορά τη σχέση μας προς τις ΗΠΑ όσον αφορά την άμυνα που προσανατολίζονται σε νέους στόχους στην εξωτερική τους πολιτική τώρα, είπα. Και έχουμε και νομοθετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά μια διαφορετική κατάσταση από τότε με το που είχαμε το πακέτο του 2009 με κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για τη δημιουργία μιας κοινή εσωτερικής αγοράς και στον τομέα της άμυνας και του αμυντικού εξοπλισμού. Αυτή είναι η γραμμή αφετηρίας, η εκκίνησης. Και εγώ θα ήθελα ουσιαστικά να πετύχω, να καταφέρουμε ότι σε όλους τους εμπλεκόμενους να καταφέρναμε, κυρίως στις κυβερνήσεις βέβαια, να πετυχαίναμε μια προσπάθεια που θα στεφόταν με επιτυχία να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση συνολικά όλοι, μια και είναι τόσο περιορισμένα τα κονδύλια πλέον και σπανίζουν. Κανονικά η βιομηχανία σίγουρα είναι ευαίσθητη στο ότι μεγαλύτερες προοπτικές, ευρύτερες προοπτικές θα έπρεπε να υπάρχουν και να διανοίγονται. Αλλά στην ειδική κατάσταση των αμυντικών βιομηχανιών που υπάρχουν πολύ λίγοι πελάτες τα ίδια τα κράτη για παράδειγμα, μια τέτοια κατάσταση είναι δυσχερής, δυσχεραίνει τα πράγματα. Και έχουμε και επιπλέον και μια κατάσταση όπου σε κάποιες χώρες, και η Σουηδία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, υπάρχουν ιδιωτικές βιομηχανίες που αντέχουν στην αγορά και είναι ανταγωνιστικές ε, και σε σχέση με άλλες χώρες όπως π.χ. στην Γαλλία έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό κρατικών τέτοιων βιομηχανιών ή εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, ώστε ας το πω έτσι, η αλληλεπίδραση μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας ε, εξοπλισμών είναι διαφορετική από ότι στη Σουηδία για παράδειγμα που είναι ιδιωτική αυτή η βιομηχανία. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη, να τα αναλύσουμε να αναλύσουμε και να δούμε πού βρισκόμαστε νομοθετικά με τις νομοθετικές προτάσεις και την υλοποίηση του πακέτου μέτρων για τα εξοπλιστικά και τον τομέα της άμυνας. Αναμένουμε να δοθούν απαντήσεις. Είναι νομίζω σημαντικό να καταφέρουμε, να πετύχουμε, να διερωτηθούμε τουλάχιστον, να ψάξουμε να βρούμε απαντήσεις πώς θα υπάρξει μια παγίωση των πραγμάτων σε σχέση και με αυτή την αγορά. Τι μπορεί να γίνει για να πετύχουμε μακροπρόθεσμα να καταφέρουμε να έχουμε ένα ισοδίκαιο, ισότιμο πεδίο δράσης, level playing field, ώστε να μπορεί η βιομηχανία μας να είναι βιώσιμη και να αντέξει. Η ανάλυση νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο. Είχαμε υπερπαραγωγή επί πολλά χρόνια. Είχαμε έλλειψη οικονομίας κλίμακας πολλά ε, διπλοεπικαλυπτόντουσαν, υπήρχαν πολλές διπλοεπικαλύψεις ε, που στρέβλωναν την κατάσταση. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό τώρα επιτέλους να δώσουμε απαντήσεις, να βρούμε απαντήσεις που μακροπρόθεσμα θα διασφαλίζουν τον χρονορίζοντα Και για την ερώτηση του Αρνό, αν σταθμίσουμε και αξιολογήσουμε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, συμπεριλαμβάνοντας ε, τον τομέα εξοπλισμών στη συμφωνία την εμπορική ΕΕ αυθόρμητα θα έλεγα ότι ουσιαστικά εκείνοι οι οποίοι είναι οι πιο ανθεκτικοί είναι οι Αμερικανοί και γι' αυτό πρέπει να μεριμνήσουμε τώρα να συνάψουμε μια τέτοια συμφωνία ή σύμβαση μαζί τους ώστε για παράδειγμα τα θέματα τροφοδότησης ε, αεροπλάνων εν πτήση να μην ρυθμίζονται, να μην αντιμετωπίζονται αυθαίρετα ή περιτροπής εκ των ενόντων και σε σχέση με τη βιομηχανία των ΙΠΑ ή την ε, γερουσία, την ε, κυβέρνηση, το σώμα, την Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν, ας το πω έτσι, κάτι το οποίο έδωσε την ευκαιρία να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν μια καλύτερη εικόνα ε, του εαυτού τους και θα ελπίζα να μπορούσαμε στο μέλλον να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο, μια καλύτερη συμβατική, ας το πω έτσι, πλαισίωση. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να το πετύχει αυτό και τι, πώς τα αξιολογεί τα πράγματα. Και είμαι πραγματικά απογοητευμένος για τα θέματα των μη επανδρομένων αεροπλάνων, αεροσκαφών, όταν βλέπει κανείς στη Γερμανία, για παράδειγμα, και το θέμα της προστασίας από τις ε, συγκρούσεις. Αλλά το πιο αποφασιστικό θέμα είναι προφανώς το ότι εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να δώσουμε την άδεια για να μπορούν να ε, λειτουργούν όλα αυτά. Εμείς ως Ευρωπαίοι μπορούμε να τα καταφέρουμε να διαπραγματευόμαστε με έναν εταίρο ο οποίος δεν μας δίνει όλες τις πληροφορίες και δεν μας αφήνει να γνωρίζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Η συνέπεια στα μη επανδρομένα αεροπλάνα είναι αυτή ακριβώς, ότι ε, χωλένουμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό όχι μόνο στα μη επανδρομένα αεροσκάφη αλλά και στους άλλους τομείς διτής χρήσης, ε, dual use για να υπάρξουν τέτοιες δυνατότητες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 να ξεκινήσουμε ώστε και στον αστικό πολιτικό τομέα και στον στρατιωτικό τομέα διτά να επιτύχουμε εκείνες τις επιπτώσεις και αποτελέσματα τα οποία χρειαζόμαστε στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για να προχωρήσουμε ως Ευρωπαίοι. Πολυάριθμα λοιπόν θέματα και ερωτηματικά αναφύονται και ελπίζω ότι από τη βιομηχανία θα έχουμε θαραλέες απαντήσεις που θα στρέφονται και θα δίνουν απαντήσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ. <coughs> Σας ευχαριστώ κύριε Κοπά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την διοργάνωση αυτής της ακρόασης και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους. Θέλω να εκφράσω την υποστήριξη της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Είναι προφανές ότι χρειάζονται μεταβολές και αλλαγές για, αλλαγές για να διευρυνθεί η βιωσιμότητα αυτού του τομέα και να υπάρξει η δυνατότητα στην οικονομική κρίση που περνάμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εκφράζοντας όμως τη θέση της ομάδας μου, δεν μπορώ όμως να αγνοήσω τις κοινωνικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν αυτές οι αλλαγές σε χιλιάδες εργαζόμενους στον τομέα. Και λαμβάνοντας αυτό υπόψη, πρότεινα όταν ε, είχαμε τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης να έχουμε και με τη συμμετοχή των συναδέλφων από την Επιτροπή Απασχόλησης και να εμπλακούν και ε, εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για να έχουμε μια ευρύτερη, πληρέστερη εικόνα και είναι πραγματικά εκπληκτικό το ότι δεν συμφώνησε το ΕΛΚ με τέτοιου είδου προτάσεις. Και γι' αυτό προτείνω το εξή ε, και θέτω το εξή. Σε ποιο βαθμό η αναδιάρθρωση τη ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων απασχόληση. Και δεδομένη τη υψηλότητα τη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, δεν θεωρείτε ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να εξεταστεί με τη μεγαλύτερη προσοχή και ποιες ε, ρήτρες ασφάλειας θα προτείνατε ή μέτρα προσαρμογής. Δεύτερη παρατήρησή μου. Συζητήσαμε σήμερα για τη βαριά βιομηχανία περισσότερο και όχι τόσο πολύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να θέτει ιδιαίτερες ε, πιεστικές ε, ε, πιέσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πώς θα μπορούσε η ιδέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη βιομηχανία να δημιουργήσει τέτοιου είδους συμμαχίες ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η βιωσιμότητά τους και ο ανταγωνισμός τους. Ποια περαιτέρω μέτρα θεωρείτε ότι θα ήταν αναγκαία και θα έπρεπε να Σα Σας ευχαριστώ. Κύριος Φανόρντεν. <clears throat> Σε ευχαριστώ. Πρώτα ζητώ συγγνώμη που έφτασα με κάποια μικρή καθυστέρηση. Άκουσα την τελευταία, το τελευταίο τμήμα της ε, παρουσίασης, αλλά όχι όλες τις ε, προηγούμενες ε, και πραγματικά ζητώ συγγνώμη για αυτή την απουσία. Σαφώς όταν κάνουμε λόγο για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Υπάρχει ένα μείγμα στόχων που εντάσσεται μέσα σε αυτή την οικονομική, βιομηχανική, στρατιωτική συνιστόσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολιτικά ένα πολιτικό επίπεδο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και γι' αυτό αυτή η ε, βιομηχανική ε, δραστηριότητα μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η πραγματικότητα όμως είναι το ότι στην αμυντική βιομηχανία τα περισσότερα γίνονται από 5-6 χώρες ε, το πολύ όλες και όλες. Εσείς περιγράψατε στην ε, Σουηδία μια επιτυχή ιδιωτική βιομηχανία που επικεντρώνεται στις αναδιόμενες αγορές και με τις ε, είπα έναν ε, εταίρο που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε. Διερωτώ με γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία και το γραφειοκρατικό της άχθος θα θέλατε να συμμετέχει σε μια τέτοια δράση. Και μια και υπάρχει ένα τέτοιο πλεονάζον δυναμικό, γιατί θα θέλατε να δημιουργήσετε ακόμα μεγαλύτερο τεχνολογικό δυναμικό, όπως φαίνεται να απορρέει από κάποια παραδείγματα που αναφέρθηκαν. Όμως φυσικά υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, συνεργασίας στην άμυνα στην Ευρώπη και είναι καλά τεκμηριωμένα αυτά και κάποια είναι επιτυχή, κάποια άλλα όχι τόσο επιτυχή. Η πιο αποτελεσματική συνεργασία είναι μεταξύ δύο εταίρων πιθανότατα και το πολύ μεταξύ τριών. Και θα σας συνιστούσα το εξαιρετικό έγγραφο από τον καθηγητή Keith Hardley και από την ε, ομάδα προβληματισμού Think Tank New Direction που έχει ε, πολύ μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτά τα θέματα. Θα σας συνιστούσα αυτή τη μελέτη. Θα έλεγα ότι ίσως ο στόχος της ε, ευρωπαϊκής ε, βιομηχανικής αμυντικής βιομηχανίας θα έπρεπε να είναι στο να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε διμερείς ή τριμερείς τέτοιες συνεργασίες ε, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε με αυτές τις ε, ε, εταιρείε, με αυτή την εταιρική σχέση όπου είναι καλύτερη αυτή γιατί στο τέλος τέλος θέλουμε να διασφαλίσουμε πρώτα ότι θα έχουμε στρατηγικά την ασφάλεια που θα ε, διατηρούμε και θα διασφαλίζουμε στις χώρες μας. Όχι σε κάποιο επίπλαστο ή μυθικό πλαίσιο, αλλά στις χώρες μας τις ίδιες συγκεκριμένα. Επ' αυτού θα ήθελα να επικεντρωθώ. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολωνικά. Επειδή εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε τον Ανόντα Ζων στην Προεδρία της Υποεπιτροπής, με πρόλαβε, έθεσα ακριβώς τις δύο ερωτήσεις που ήθελα να θέσω εγώ. Δηλαδή, την ερώτηση σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ μα σχέσει στην ε, διαπραγματεύσει ελεύθερων συναλλαγών με τι ΗΠΑ και τη δεύτερη μου ερώτηση για τα ντρόν, τα μη επαδρομένα αεροσκάφη. Με πρόλαβε και στι δύο ερωτήσει, γιατί πραγματικά αυτά τα δύο θέματα είναι εξαιρετικά σημαντικά για μας. Για το θέμα λοιπόν της συνεργασία με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουμε πάρα πολλού ε, δεσμού ε, μεταξύ των, ευρωπαϊκών και των αμερικανικών εταιριών. 30.000 ε, ε, ε, απασχολούνται Ευρωπαίοι σε αμερικανικές εταιρείες. Επίσης έχουμε και στην Πολωνία τα Augusta Westland και έχουμε και υφιστάμενθα και τον αμερικανικό ανταγωνισμό για την κατασκευή τέτοιων ελικοπτέρων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και δεσμών και σχέσεων λοιπόν με τις Ηνωμένε Πολιτείες στα θέματα εμπορίου. Αλλά έχω να θέσω και μια άλλη ερώτηση πολλοί εμπειρογνώμονες είπαν ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ευρώπη γενικώ κατασκευάζονται ε, πολλά αεροσκάφη που θα θέλαμε να πουλήσουμε και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε γενικώ ε, υπερπαραγωγή αμυντικού εξοπλισμού κατασκευάζουμε και τεθωρακισμένα και πολλά ελικόπτερα. Έχουμε και πολλά ναυπηγεία που κατασκευάζουν πολεμικά πλοία. Πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνουν συγχωνεύσεις τέτοιων μεγάλων μονάδων παραγωγής ή θα οδηγηθούν ορισμένες αναπόφευκτα στο κλείσιμο γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι βιομηχανίες για τις χώρες μας και τις πόλεις μας, γιατί απασχολούν ε, πολλούς εργαζόμενους. Ευχαριστώ. merci Ευχαριστώ. Πριν ακούσουμε τις απαντήσεις από τους ε, βιομηχανούς, ο κύριος Νιούλιν. Ίσως ε, μετά από όσα άκουσες από τους ομιλητές, ή τις ερωτήσεις ε, να έχει τροποποιήσει λιγάκι τα όσα σκόπευε να πει. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω εν συντομία αυτό που έκανα εγώ και τρεις από τους συναδέλφους μου για τους τελευταίους τρεις μήνες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ετοιμάσαμε μία μελέτη για την τρέχουσα κατάσταση και, την, και το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας ο Μπαλέρο Μπαϊάνι, ο Ιταλός, ο κ. Βάλασεκ επίσης, ο οποίος άλλαξε δουλειά. Ε, τι κάναμε λοιπόν το τελευταίο διάστημα. Εξετάσαμε το θέμα αν υπάρχει η ευρωπαϊκή τεχνολογική βιομηχανική αμυντική βάση. Θέλω να έχετε ξεκάθαρο τουλάχιστον αυτό το θέμα όταν τελειώσει η σημερινή συνεδρίαση. Το θέμα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε την προμήθεια του αμυντικού υλικού και των υπηρεσιών απέναντι σε πολιτικούς κινδύνους γιατί, ας πούμε, μπορεί ε, οι γειτονές σας να μην ε, επιτρέπουν την διέλευση αυτών των, ε, αυτού του εξοπλισμού, ας πούμε, μέσα από τα σύνορά τους κτλ. Ε, είχε η χώρα ή οι ένοπλες δυνάμεις σας αυτά τα, αυτό το υλικό στη διάθεσή της. Τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Η αλυσίδα παραγωγής είναι όλο και πιο διεθνής εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο εθνικός ανεφοδιασμός και η ασφάλεια του ανεφοδιασμού είναι μύθος. Του αρέσουν, αρέσκουν τα κράτη-μέλη να μιλάνε γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή η ιδέα έχει εξαλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το 2007 τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ε, συμφώνησαν για αυτή τη στρατηγική EDTIB ε, που δημιουργήθηκε για να μειώσει τις πιέσεις ανάμεσα στην πολιτική και βιομηχανική δυναμική. Και αυτό που συνέβη σήμερα είναι ότι έχουμε χάσει ε, περίπου μισή δεκαετία. Ε, η EDTIB στην Ευρώπη μειώνεται, οι εθνικές στο βαθμό που υπάρχουν ε, αυξάνονται λιγάκι, αυτή η αμυντική βάση δηλαδή, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη την ευρωπαϊκή διάσταση. Έχουμε μια συνεχή εθνικοποίηση στην αμυντική βιομηχανία και έχουμε από την άλλη όμως αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση στον πλανήτη. Επομένως, το αποτέλεσμα της μελέτης μας είναι ότι χρειαζόμαστε μία αντίστροφη προσέγγιση στην, στους αμυντικούς βιομηχανικούς στόχους και μέσα. Πρέπει να αξιολογήσουμε τι μπορούμε να πετύχουμε ως Ευρώπη ή μήπως πρέπει να αλλάξουμε τελείως αυτή την προσέγγιση, το EDTIB, την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Βιομηχανική Αμυντική Βάση. Αυτή η αμυντική βάση δημιουργήθηκε γιατί ο, η ασφάλεια του εθνικού ανεφοδιασμού δεν ήταν πλέον βιώσιμη ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να πληρώσουμε πια για αυτήν. Και θα πρέπει να εξασφαλιστεί στα κράτη-μέλη η δυνατότητα ότι έχουν το αμυντικό υλικό που χρειάζονται, αλλά θα πρέπει να περάσουν από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή ήταν η ιδέα. Ε, η ιδέα ήταν αυτή, ήταν ένα πολιτικό όραμα, μια θεώρηση ότι ας πούμε, θα πρέπει το πολιτικό και το βιομηχανικό επίπεδο της Ευρώπης κάπου να συγκλίνουν. Το ένα να ακολουθεί το άλλο. Αυτό στα μέσα της ε, δεκαετίας του 2000. Αριστερά βλέπετε το πολιτικό όραμα και κάτω δεξιά βλέπετε ε, ποια ήταν η Ευρώπη το 2007. Ότι υπήρχε ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό και το εθνικό EDTIB. Να μην αυτή βάση. Ε, υπάρχουν δηλαδή παράλληλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν συνδέονται. Δεν συνδεόταν, εν το 2007. Πώ αναγνωρίζουμε αυτή την αμυντική βάση όταν τη βλέπουμε, Ε, το EDTIB ε, που υπάρχει στην Ευρώπη δεν είναι το αποτέλεσμα, το άθροισμα των εθνικών συνιστοσών. Είναι η διαφορά. Ε, κανονισμοί, πολιτικές που ενισχύουν την ε, ευρωπαϊκή διάσταση μέσω της βιομηχανίας. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο ανταγωνιστική από ότι αν συγκριθεί αυτή με τις εθνικές ε, αμυντικές βιομηχανίες. Επίσης, ε, να, εξαρτήσουμε, να μειώσουμε και την εξάρτηση από παράγοντες και χώρες εκτός Ευρώπης. Στο διεθνές επίπεδο, έχουμε κλασικές ε, συνήθειες για συνεργασία που υπάρχουν. Έχουμε το άρθρο 346 που ε, επινοήθηκε δεκαετίες πριν το παλιό άρθρο 223 που άλλαξε νούμερο, αλλά επιβίωσε σε όλες τις ευρωπαϊκές εφαρμογές. Ε, αυτό σε σύγκριση με τον διακυβερνητικό τρόπο ε, συνεργασίας, είχαμε ένα πολλαπλασιασμό θεσμικών οργάνων, έχουμε την Κομισιόν, έχουμε την ΕΝΤΑ, έχουμε την ε, Συνθήκη της Λισαβόνας, στην Κομισιόν, αλλά καμία επίπτωση όλων αυτών στην πολιτική μέχρι σήμερα. Σε πολιτικό επίπεδο, σε εθνικό, και σε εθνικό επίπεδο, ε, η κατάσταση που υπάρχει εξηγεί γιατί δεν γίνεται τίποτα σε διεθνέ επίπεδο. Έχουμε τα κράτη LOL, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και βάζουμε και την Πολωνία, γιατί είναι ανερχόμενος παίχτης. Αυτές οι 6-7 χώρες είναι το 20% των ευρωπαϊκών κρατών ή το 80% του προϋπολογισμού. 81 δισεκατομμύρια είναι ο κύκλος εργασιών. Αυτές οι 6-7 χώρες τέλος πάντων, η, πολίτια, η πολιτική προμηθειών, ε, πολιτική αγοράς δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Οι εθνικές επιρροές διατηρούνται στο βαθμό του δυνατού και αυτό επηρεάζει και την εθνική δομή της αμυντικής βιομηχανίας. Θα επανέλθω σε αυτό και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει. Γενικά σημαίνει ότι οι παραγωγοί αγοράζουν εσωτερικά ε, τα τεθωρακισμένα, τα αεροπλάνα, τα νεαρία οχήματα, τα σκάφη, τα αγοράζουν εσωτερικά. Η μη παραγωγή αυτοί που δεν έχουν δηλαδή μεγάλη αμυντική βιομηχανία εσωτερικά, δεν ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν αγοράζουν στην Ευρώπη, αγοράζουν όπου τους βολεύει. Ε, το JSF, το πρόγραμμα αυτό, βλέπετε το πρόγραμμα των F-16, επομένως δεν μετράει εδώ η Ευρώπη. Και για το μέλλον, ε, η πρόγευση που έχουμε, έχουμε δηλαδή μείωση των πολυεθνικών προγραμμάτων, υπάρχουν λιγότερα δηλαδή πολυεθνικά προγράμματα, υπάρχουν περισσότερα διακρατικά, διμερεί αν θέλετε, ή εθνικά και κυρίως τα, δι, τα διμερεί αυτά είναι διατλαντικά. Έχουμε λιγότερες προμήθειες. Έχουμε δηλαδή μεταφορά ε, των προμηθειών στην προσφορά. Ε, συντήρηση, διατήρηση. Άρα η, η ιστορία που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι υπηρεσίες και όχι οι προμήθειες στον αμυντικό τομέα. Τώρα, Έχουμε τέσσερα διαφορετικά τμήματα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανία, αεροναυπηγική, ε, χερσαίας τομέας, ναυτικός τομέας και ηλεκτρονικά. Ε, η αεροναυπηγική είναι ο μεγαλύτερο τομέα ε, και υπάρχουν βασικέ διαρρέσει από του τέσσερι τομεί. ο τομέα των ηλεκτρονικών και τη αεροναυπηγική και οι εταιρείε σε αυτόν τομέα, σε αυτούς τους τομέες, εξαρτώνται λιγότερο από τις αμυντικές δουλειές, από τις τους άλλους τομείς. Παραδείγματο χάρη στον χερσαίο και θαλάσσιο τομέα, ε, έχουμε εξειδικευμένες εταιρείε στην Ευρώπη που εξαρτώνται από τα έσοδα που έχει ο στρατιωτικός κλάδος, από τα κονδύλια που έχει στη διάθεσή του. Το βλέπετε αυτό και στα προγράμματα και στη συνεργασία. Ο τομέας ενοπηγικής είναι πάρα πολύ θεσμοθετημένος. Έχουμε δηλαδή ε, σαφώς ε, πολύ εθνικά προγράμματα και εταιρείε, σαφώς προσδιορισμένα, ενώ στους άλλους τομείς, ε, χερσαίο και θαλάσσιο, συνεργασία δεν υπάρχει τόσο συχνά και δεν είναι πολύ επίσημη, θεσμοθετημένη κτλ. Για να δούμε διαφορετικά την ε, βιομηχανική Ευρώπη. Οι βασικές ε, εταιρείε, ε, η ΜΠΑΕ, η ΕΝΤΑΣ, η Θάλες, η Φινμεκάνικα, είναι παγκόσμιοι εταίροι, δηλαδή τα περισσότερα χρήματά τους τα βγάζουν από αλλού από τον κόσμο, όχι κατά από την Ευρώπη. Και έχουμε μια συγκέντρωση των πέντε μεγαλύτερων εταιριών στην Ευρώπη, όπου τα δύο τρίτα των, του κύκλου εργασιών τους ισούνται με τον υπόλοιπων 40 μεγάλων εταιριών. Έχουμε κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, όπου έχουμε τις μεγάλες εταιρείες, ε, και στην Ανατολική Ευρώπη έχουμε μικρές εταιρείες, ε, με εξαίρεση μία-δύο. Δηλαδή έχουμε μία ε, περιφερειακή ανισορροπία. Αν δείτε και τους τομείς, βλέπετε ότι η ενοποίηση στον τομέα των θαλάσσιων και χερσαίων και χερσαίων τομέα έχει προσκρούει πάρα πολλά εθνικά εμπόρια. Υπάρχουν αυτές οι εταιρείε, αλλά δεν μπορούν να ενισχυθούν περισσότερο, να ενοποιηθούν περισσότερο, γιατί τις προστατεύουν οι κυβερνήσεις τους, ε, οι οποίες θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εταιρείε τα επόμενα χρόνια ή για τα επόμενα προγράμματα. Προσπαθώ να εξηγήσω τώρα αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο εδώ σε εσά. Ε, εδώ έχουμε τους τέσσερις τομείς. Πάνω δεξιά και κάτω αριστερά έχουμε τον ε, χερσαίο και θαλάσσιο τομέα και οι μεγάλες ε, χριστουγεννιάτικες μπάλε. Εκεί έχουμε το 100% των εταιριών που είναι ενεργές σε αυτούς τους τομείς μόνο. Και έχουμε πέντε εταιρείε στο θαλάσσιο τομέα που, παίρνουν, που βγάζουν χρήματα μόνο από εκεί, από το θαλάσσιο τομέα δηλαδή. Δηλαδή δεν έχουν ε, άλλους τομείς, τους υπόλοιπους τρεις. Δηλαδή αν δεν πάρουν λεφτά από τις θαλάσσιες ε, δουλειές ας πούμε, κλείνουν. Επίσης, στα χερσαία συστήματα έχουμε λίγες εταιρείες ε, εξειδικευμένες που έχουν μόνο τέτοια συστήματα και δεν έχουν πουθενά αλλού εμπορικά, μη στρατιωτικά, εν πάση περιπτώσει, στρατιωτικές δραστηριότητες, είτε στο, στην αεροναυπηγική, είτε στα ηλεκτρονικά, είτε αλλού. Δεν έχουν. Επομένως, έχουμε αυτή την τάση ε, τελείως διαφορετική από ό,τι συμβαίνει στους άλλους δύο τομείς, ηλεκτρονική ας πούμε και αεροναυπηγική. Εκεί σχεδόν καμία εταιρεία δεν εξειδικεύεται αποκλειστικά στα ηλεκτρονικά ή στην αεροναυπηγική. Έχουν δραστηριοποιούνται σε πολλούς κλάδους, δεν υπάρχει εξειδίκευση και συχνά ε, έχουν και, κάνουν και δουλειά στον εμπορικό, μη στρατιωτικό δηλαδή τομέα. Επίσης, έτσι για να σας δώσω ένα δύο πράγματα, οι μεγάλες μπλε μπάλες που είναι τα συστήματα BAE. Σχεδόν 100% ε, εκτός από τα λεωφορεία που φτιάχνουν για τις Ηνωμένες συγγνώμη, για το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, βγάζουν τα λεφτά τους σχεδόν 100% δηλαδή από το στρατιωτικό τομέα. Ε, και τα πάνε και στους τέσσερις ταμείς πάρα πολύ καλά. και για τη Φινμεκάνικα και για το Θαλή, το Τάλες, είναι το, ισχύει το ίδιο σε σχέση με άλλες εταιρείε που είναι εξειδικευμένες και εθνικές και που ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε δηλαδή αυτούς τους δύο ακραίους πόλους που υπάρχουν ε, στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Το σημαντικό πράγμα στο EDTRB ήταν, αρχικά ήταν οι εξαρτήσεις, η στρατιωτική εξάρτηση, δηλαδή εξάρτηση από η Ρωσία, από τους Αμερικανούς, από προμηθευτές ξένους, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μειωθεί. Αυτό είναι καλό. Το κακό ποιο είναι, και δεν το ξέρουν τα κράτη-μέλη, ότι έχουν αποκτήσει νέες μορφές, ιδίω βιομηχανική εξάρτηση έχει αποκτήσει αυτή η εξάρτηση. Νέα μορφή εξάρτησης λοιπόν έχει. Προσπαθούμε να καταλάβουμε κάθε φορά τι είναι η εξάρτηση ε, παραδείγματος χάρη για τους, η Τοσίμπα παράγει ημιαγωγούς. Δεν ε, εδρεύει στην Ευρώπη, αλλά στην Ταϊλάνδη, στην Ασία, που είναι ο μόνος τόπος παραγωγής ημιαγωγών για τους κλούς δίσκους. Δεξιά βλέπετε την Ταϊλάνδη το 2011, είχε πλημμυρίσει και σταμάτησε η παραγωγή ημιαγωγών σκληρών δίσκων εντελώς για όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή για μη ε, στρατιωτική χρήση, αλλά και για τη στρατιωτική χρήση. Είναι μια εξάρτηση που υπάρχει και δεν είναι ευρωπαϊκή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτή. Ε, γιατί ούτω ή άλλω δεν έχουμε πια κέντρα παραγωγή στην Ευρώπη. Πουθενά. Υπάρχουν πολλέ άλλε αντίστοιχε εξαρτήσει. Μπορεί να εξαρτάσει από υλικά, α πούμε. Παραδείγματο χάρη, στα πολεμοφόδια η Ευρώπη εξαρτάται από, α, ε, από την Κίνα για λευκό φόσφορο. Για να παράγουμε τα πυρομαχικά μας. Αυτό είναι μια, μια άλλη πλευρά της εξάρτησης. Ε, χρειαζόμαστε να εισάγουμε όλα αυτά τα υλικά. Επίσης εξαρτώμαστε, εξαρτώμαστε και στις εξαγωγές. Δηλαδή, αλλιώς οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βγάλουν τζίρο. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βγάζουν τα λεφτά τους εκτός Ευρώπης. Επομένως, για να επιβιώσουν θα πρέπει να εξάγουν εκτός Ευρώπης. Και σε αυτόν τον τομέα, λοιπόν, η Ευρώπη δεν μετράει πια για την αμυντική βιομηχανία. Για να τελειώσω με αυτή την ανάλυση, το μέλλον της ευρωπαϊκής EDTIB ε, είναι το ίδιο με ό,τι ήταν τα τελευταία πέντε χρόνια, συνεχιζόμενη εθνικοποίηση, αύξηση της ε, παγκοσμιοποίησης. Η EDTIB συνδέεται με πολλά δρόμενα εκτός Ευρώπης, παρά με αυτά που συμβαίνουν εντός Ευρώπης. Έχουμε, έχουμε μια μεγάλη ε, ξένη η DTIB. Ε, στην Ευρώπη μειώνεται. Οι συστάσεις μετά από όλα αυτά. Η πρώτη σύσταση δεν, αφορά, δεν απευθύνεται προς τα κράτη-μέλη, αλλά τους πελάτες, που τώρα είναι τα κράτη-μέλη βέβαια. Αν θέλουν ασφάλεια του εθνικού ενεφοδιασμού, ασφάλεια του εθνικού ανεφοδιασμού πρέπει να, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει πια εθνικό ανεφοδιασμό, πρέπει να είναι ευρωπαϊκό ανεφοδιασμό και άρα θα πρέπει να αναθεωρήσουν τη στρατηγική του. Δεν μπορούν πλέον σήμερα να βασίσουν στρατηγική του 2007. Επίση, χρειάζεται μια συνεχή πολιτική δέσμευση να υπερασπιστούν τη βιομηχανία αυτή. Στο τελευταίο συμβούλιο που συζητήθηκε η άμυνα ήταν το 2008. Και τώρα θα γίνει ένα ακόμα Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται ετήσια τέτοιου τύπου συζητήσει σε επίπεδο Συμβουλίου και δεν θα πρέπει να ασχολείται το Συμβούλιο μόνο με την αμυντική βιομηχανία, αλλά με την άμυνα αυτή καυτή. Επίσης, αυτό που είναι αναγκαίο είναι αυτό που κάναμε προς το παρόν, μια φορά παρακολούθηση δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην ευρωπαϊκή τεχνολογική βιομηχανική αμυντική βάση. Γιατί η εντύπωσή μου είναι ότι ούτε η Κομισιόν ούτε η ΕΝΤΑ έχουν σαφή εικόνα για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Και δεν είναι σωστή η βάση αυτή για να δημιουργήσουμε, να προκύψουν συστάσεις για το Συμβούλιο Άμυνας αυτή. Κάτι άλλο. Η διαδικασία. Αν θέλουμε να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική ή να να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο. Το θέμα δεν είναι μόνο να εφαρμόσουμε αυτά που μας λένε τα κρατημέλη Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση και διάγνωση της κατάστασης. Στη συνέχεια θα προβούμε σε μεταρρύθμιση των στόχων και των μέσων. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε δηλαδή τη σωστή ε, σειρά. Επίσης η στρατηγή είναι ένα κύκλου. Θα πρέπει να γίνεται τακτικά αξιολόγηση το κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι στόχοι, μια και μια φορά το χρόνο ίσως. Αλλιώς θα επαναρχόμαστε μετά από πέντε χρόνια και δεν θα έχουμε καν τη δυνατότητα να μιλούμε για ευρωπαϊκή τεχνολογική βιομηχανική βάση στον τομέα άμυνας και ασφάλειας. Ευχαριστώ. Στην παρουσίασή σας ε, βρήκαμε και κάποια σημεία που είχαν προαναφέρει οι καλεσμένοι μας στις δικές του ομιλίες. Για παράδειγμα, το θέμα το ότι δεν έγινε μια παρακολούθηση, εξολόγηση των προηγούμενων αποφάσεων σε διαφορά τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Βιομηχανική Βάση ή για την ε, οδηγία για το αμυντικό πακέτο. Βέβαια, η μετάθεση στις, τεχνικές, στις εθνικές ομοθεσίες έγινε με κάποια καθυστέρηση. Αλλά δεν ε, αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος αυτών των νομοθετικών διατάξεων ε, στην αμυντική βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητά της. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους ε, ευρωβουλευτές και στους καλεσμένους μας. Πρώτα στους καλεσμένους ε, με αντίστροφη σειρά. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιάνν Πι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολλές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω κάποιες, ε, τουλάχιστον και εκείνες του κυρίου Φανόρντεν. Αυτό που προσπαθώ να πω κυρίως είναι το ότι πιστεύουμε υπό την εμπειρία και προοπτική της Σουηδίας ότι πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά μας στην Ευρώπη και οι συνήθειές μας όσον αφορά τις προμήθειες στην Ευρώπη πάνω από 80% γίνονται σε εθνική βάση κυρίως. Είναι πολύ κλειστή η ευρωπαϊκή αγορά και ο λόγος για τις σουηδικές εταιρείες που επικεντρώνονται όλο και περισσότερο προς τις ΗΠΑ και στις ε, αναδιόμενες αγορές είναι ότι έχουν προβλήματα να έχουν πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τη νέα οδηγία για τις ε, προμήθειες ε, και τις αγορές εξοπλιστικού υλικού και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με το, την χρήση του αντίστοιχου άρθρου με το δυνατόν πιο αυστηρό πλαίσιο και να είναι το δυνατόν πιο περιορισμένες οι εξαιρέσεις διότι θέλουμε να υπάρχει ανοιχτός ανταγωνισμός στο μέτρο που μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Αυτό ήθελα να πω στην παρουσίασή μου. Και όσον αφορά τις συμπράξεις, clusters και κέντρα υπεροχής, ε, centers of excellence, αν υπάρχει, υπάρχουν κονδύλια για τέτοια προενταχθέντα ε, κέντρα υπεροχής. Αν δεν υπάρχουν τότε καλύτερα να παραμείνουμε σε έναν μηχανισμό γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε ανταγωνιστική σύμπραξη. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι μια δυναμική σύμπραξη και να δούμε πώς θα πετύχουμε αυτή τη δυνατότητα συμμετοχής και συνεργασίας. Αυτό πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν προκαθορίσουμε πού θα πάνε τα κονδύλια και έχουμε απλά και μόνο κάποιους που θα μεριμνούν για την εφαρμογή αυτών, δεν θα έχουμε ε, προώθηση του ανταγωνισμού και ένα ανοιχτότερο πλαίσιο. Αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αν θέλουμε να συνεργαστούμε πρέπει να γίνεται με διμερή ή τριμερή ε, μορφή. Όσο περισσότερες χώρες συμμετέχουν τόσο μεγαλύτερα τα προβλήματα και τόσο πιο περίπλοκος ο χαρακτήρας ε, αυτών των προγραμμάτων. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 5, 6, 10, 12 κράτη που θα συμμετέχουν. Θα πρέπει όμως ε, να είναι ανοιχτή η δυνατότητα για τις βιομηχανίες της Ευρώπης ε, να μπορούν να συμμετάσχουν. Αυτό είναι υπό τη δική μου προοπτική μια απάντηση που θα θέλαμε να δώσουμε σε μια άλλη ερώτηση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πιστεύω και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε πολύ και σε βάθος στη Σουηδία όταν η Σουηδική Βούλη ε, ανέφερε το ότι θα είχαμε μείωση των προμηθειών και θα φοβόμαστε ότι θα είχαμε απώλεια θέσεων απασχόλησης και αυτό που ε, θελήσαμε να πετύχουμε είναι να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Ένα καλός τρόπος λοιπόν είναι, αν θέλουμε να απολεστούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, να συνεχίσουμε όπως ε, μέχρι σήμερα. Θα πρέπει μόνο ανοίγοντας τον ανταγωνισμό να δούμε ότι υπάρχει μια προοπτική να υπάρξει βελτίωση με τη συμμετοχή και πρόσβαση εταιριών στην ε, αγορά, ευρωπαϊκή αγορά. Δεν λέω ότι θα διασφαλιστούν και θα μείνουν οι θέσει απασχόληση στου ίδιου βιομηχανικού κλάδου όπω σήμερα. Είμαι υπέρ του να εξετάσουμε και να δούμε πώ θα μπορούσαν περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, να δραστηριοποιούνται σε περισσότερε χώρε. Αλλά πρέπει να υπάρχει αναγνώριση για να γίνει αυτό τη πρόσβαση ε, στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ή δεδομένο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρωμητή. Ευχαριστώ. Εγώ φυσικά θα αναφερθώ κυρίως στην αγορά ελικοπτέρων και το θέμα της στήριξης της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, γιατί θεωρώ ότι η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και αυτού του κλάδου και γενικώ της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας εξαρτάται από την ε, ικανότητα να προσφέρουν πραγματικά πρωτοπόρα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Και όπως είπε και προηγουμένως ε, στην ομιλία μου, αυτό μπορεί να γίνει είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων, όπως ε, είχαμε το αμερικανικό μοντέλο, με αναφέρθηκε το GMR, ένα πρόγραμμα της ε, Αμερικανικής ε, Άμυνας, που περιλαμβάνει ε, και ένα σημαντικό σκέλος άμυνας, έρευνα, συγγνώμη, γιατί μιλάει για μεταφορές υψηλής ταχύτητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθετης απογείωσης και προσγείωσης ή μπορούμε να έχουμε κέντρα αριστείας και πόλους συγκεκριμένους κλάστερς με ειδίκευση συγκεκριμένη. Επίσης και στο θέμα των δαπανών θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αμυντική βιομηχανία χάρη σε μεγαλύτερο εξορθολογισμό της εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Και στη δική μας περίπτωση μιλήσαμε για τη χρήση των πλατφορμών, είτε σε στρατιωτικό είτε στον πολιτικό κλάδο. Και χάρη σε αυτές τις πλατφόρμες θα έχουμε καλύτερη απόσβεση του κόστους ανάπτυξης ενός μοντέλου και θα έχουμε χαμηλότερο κόστος εμπορευματοποίησης. Κάτι άλλο που χρειαζόμαστε είναι η υποστήριξη σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές μας. Γιατί έχουμε το αντίθετο παράδειγμα της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί έχουμε το FMS ή άλλους περιορισμούς εισαγωγικούς εξαιτίας της νομοθεσίας ΙΤΑΡ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, και είχαμε και το αντίθετο παράδειγμα της μη πρόσβασης τέτοιων μηχανισμών όταν μιλούμε για κάποια μέσα προστασίας. Η βιομηχανία λοιπόν κατασκευής ελικοπτέρων έχει προχωρήσει πολύ, έχει συμβιώσει μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά τι συγχωνεύσει, τι συνεργασίε. Είχαμε την χαρακτηριστική συγχώνευση Augusta Westland και τη συγχώνευση τριών βιομηχανιών πολωνικής, ιταλικής και Βρετανικής βιομηχανίας και είχαμε και αντίστοιχη συγχώνευση Ισπανικής, Γερμανικής και Γαλλικής ε, βιομηχανίας. Ήταν ε, ε, συγχωνεύσει αρκετά περίπλοκες, αλλά σίγουρα επιθυμητές και ζητούμενο ήταν η εξισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων περιοχών και αξιοποίηση της αριστείας που είχε η κάθε βιομηχανία στον κλάδο της μπορούμε να αποφύγουμε, πιστεύω, τις επικαλύψεις και στον τομέα της προσφοράς. Καλό θα ήταν λοιπόν να βαθύνουμε και στο θέμα αυτό. Αυτά για το δικό μου κλάδο τουλάχιστον. Και ο κύριος Τραπιέ τώρα. Τώρα, για την αεροναυπηγική βιομηχανία, εγώ θα μιλήσω περισσότερο για τα ντρόνα, αυτά τα μη επαδρομένα αεροσκάφη, γιατί υπευλήθησαν πολλές ερωτήσεις. Όταν η Ευρώπη συνενώνεται και συμμαχεί, όταν ε, γίνονται διάφορες συμμαχίες, ε, ε, μεγαλουργεί πραγματικά η Ευρώπη. Είχαμε την περίπτωση Γαλλίας, Ιταλίας, Σουηδίας, Ισπανίας, Ελλάδας και Ελβετίας που συνεργάστηκαν για την κατασκευή ενός μαχητικού ντρόν 400 εκατομμύρια ευρώ και είμαστε απαιτητικοί παρά τα ισχνά κονδύλια. Οι Αμερικανοί ξοδεύουν πολύ περισσότερα και παρόλα αυτά είμαστε ε, και ανταγωνιστικοί και έχουμε και τον προπολογισμό για αυτό. Όχι υπερβολικό, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και με τις έξι αυτές χώρες, με τις έξι βιομηχανίες, έχουμε καταρτήσει κανόνες με βάση τους οποίους κάθε βιομηχανία που προσφέρει μια τεχνολογία ή που την αναπτύσσει κρατά την κυριότητα αυτής της ε, βιομηχανίας, αυτού του του, της βιομηχανίας και μπορεί να τη θέσει για κοινή χρήση με σεβασμό όμως της πνευματικής ιδιοκτησίας, των πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλαδή τα, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις παροχής αυτής της τεχνολογίας θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα της αγοράς, το εμπορικό δηλαδή. Και αυτό συζητούμε και στα πλαίσια της, ε, του ορίζοντα 2020. Υπάρχουν δυνατότητες λοιπόν για κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μη επαδρομένα αεροσκάφη επιτήρησης. Ε, εδώ και καιρό η βιομηχανία και μάλιστα έχουμε και διάφορες ομάδες σκέψης. Ε, στην ΑΕΣΤ έχουμε το Aircraft Sectorial Group, έχουμε την RDS, Filmechanica, sub Dassault, σε αυτή την Ένωση Αεροναυπηγικής Διαστήματος και Άμυνας και στις ομάδες αυτές ε, προβληματισόμαστε από κοινού για τα θέματα αυτά. Και εδώ και 15 χρόνια προσφέρουμε στις αρχές μας, είτε στις εθνικές είτε στις ευρωπαϊκές, ε, ε, κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για μια επανδρομένα αεροσκάφη και στην Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ε, κάνουμε την πρόταση Fast for Europe ε, με την υπογραφή όλων των ε, βιομηχάνων που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Οι βιομήχανοι λοιπόν ανέλαβαν τις ευθύνες τους και αν αύριο εφαρμόσουμε το pooling and sharing, αυτή τη συνένωση και την κοινή χρήση για τα καταδιοκτικά στην Ευρώπη, θα έχουμε ένα δεύτερο FM35. Τώρα, στην ε, Γαλλία έχουμε και 100% ιδιωτικές επιχειρήσεις και πάνω από το 80% του κύκλου εργασιών τους γίνεται στο πολιτικό τομέα και όλο και λιγότερο στο στρατιωτικό. Το ίδιο ισχύει και για την ε, ΑΕΣΔ, την Ένωση αυτή Αεροναυπηγικής Διαστήματος και Άμυνας. Και τα περισσότερα χρήματα τα βγάζουν από πολιτικά ελικόπτερα. Είναι θέμα πολιτική λοιπόν. Θέλουμε να κρατήσουμε, να διαφυλάξουμε τεχνολογίε που συμμετέχουν στην άμυνα στην Ευρώπη και συμβάλλουν στην άμυνα. Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είχαμε ανταγωνιστική παραγωγή. Αν όμω θέλουμε να συγκριθούμε με τα αμερικανικά προϊόντα που ήδη έχουν, βρίσκονται σε, σε μεγάλο στάδιο ανάπτυξη και έχουν καταβροχθήσει δισεκατομμύρια δολάρια και εμεί πρέπει να αποσβέσουμε τα εκατοντάδε εκατομμύρια και όχι τα δισεκατομμύρια υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα. Γι' αυτό και λέω ότι στην οδηγία θα πρέπει να, είμαστε, να έχουμε πραγματικέ πραγματικές συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και να υπάρχει και μια συγκρισιμότητα. Αν οι χώρε εκτό Ευρώπης αφενός ε, ε, επενδύουν μαζικά στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ εμείς ε, έχουμε ισχυρές επενδύσει, όσο και αν συνεννόμαστε και συνεργαζόμαστε, θα βρεθούμε σε δυσμενή θέση. Και ειδικά οι ιδιωτικέ επιχειρήσει θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και θα επικεντρωθούν περισσότερο στο μη στρατιωτικό κλάδο. Παράδειγμα, η Airbus. Και θα προσανατολιστεί σε άλλου τομεί, μακριά από το στρατιωτικό. Είναι θέμα πολιτική επιλογή λοιπόν. Τι θέλει η Ευρώπη για τη βιομηχανία τη. Και το είπαμε και προηγουμένως, θα υπάρξει και βιομηχανικός αντίκτυπος και κοινωνικός αντίκτυπος από τις επιλογές αυτές, γιατί ο μη στρατιωτικό τομέα, για να επιβιώσει απέναντι στην ανταγωνιστικότητα των αδειωμένων οικονομιών και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που επαναλαμβάνω παράγει σε δολάρια, θα πρέπει να κάνει να μετεγκαταστάσει, να μετεγκαταστήσει τις επιχειρήσεις της. Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο με βάση τα όσα είχαμε προβλέψει. Ορισμένοι από εσά έχουν επιπλέον παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Ας επωφεληθούμε από την παρουσία των ομιλητών μας. Μήπως, βλέπω οι ευρωβουλευτέ δεν θέλουν να προσθέσουν κάτι, μήπως κάποιο ομιλητή, κάποιο από το πάνελ θέλει να προσθέσει κάτι, ο κύριος Μέρλινγκ. Ναι. Δύο πράγματα θέλω να πω. Κάτι που παραβλέπεται και στη χώρα μου. Ε, η αμυντική βιομηχανία προσφέρει και θέσεις απασχόλησης. Ε, στο, την εποχή του ψυχρού πολέμου ήταν πολύ α, ισχυρός τομέας. Ε, οι δουλειές τώρα, οι θέσεις απασχόλησης ε, που εξαρτώνται από το αμυντικό ε, τομέα είναι ε, περίπου 500.000. Ε, είναι 0,024% όλων των ε, θέσεων. Δεν ε, μετράει, δηλαδή, με την έννοια των θέσεων απασχόλησης, αλλά μετράει γιατί είναι στρατηγικός τομέας. Νομίζω η βιομηχανία θα πρέπει να προβάλλει αυτό το επιχείρημα, ότι είναι στρατηγική σημασία και όχι τόσο ότι δίνει θέσεις απασχόλησης. Χρειαζόμαστε αυτή η βιομηχανία γιατί είναι στρατηγικά σημαντική. Γιατί δεν θέλουμε να εξαρτώμαστε από άλλους. Όχι γιατί ε, το, ο κύκλος εργασιών είναι πολύ σημαντικός. Ούτως ή άλλως είναι, αν το θέσουμε οικονομικούς όρους, είναι κρατικοδίαιτος τομέας. Τώρα για την εξάρτηση. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα αν δεν υποστηρίξουμε αυτή τη βιομηχανία, τα επόμενα 20 χρόνια θα εξαρτηθούμε από άλλους. Μέχρι να φτάσουν τα νέα προγράμματα. Οι κάποιες νέες βιομηχανίες θα εξαφανιστούν. Και ποιοι θα εξαφανιστούν, ποιοι θα διατηρηθούν, είναι ποιοι θα πάρουν το θέμα είναι ποιοι θα πάρουν δηλαδή, τις περισσότερες κρατικές επιδοτήσεις ή ποιοι είναι πιο ανταγωνιστικοί. Έτσι θα παιχθεί το παιχνίδι. Επίσης, βασικό είναι, ε, ωραία, θα, δεν θα μπορούμε να βασιστούμε στη δική μας ε, αμυντική βιομηχανία. Σε ποιου θα βασιστούμε. Θα εξαρτηθούμε ε, από τους ε, Κινέζους, τους Κορεάτες. Μάλιστα. Κρατάμε αυτές τις δύο παρατηρήσεις που συγκλίνουν κιόλας και επανεπιβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για ένα τομέα πολύ πολιτικό, που υφίσταται δηλαδή τις συνέπειες των πολιτικών αποφάσεων πολύ περισσότερο από άλλους οικονομικούς τομείς. Εξού και η ιδιαιτερότητα της αμυντικής βιομηχανίας. Μια ιδιαιτερότητα, για να το πω ειλικρινά, που δεν ελειφθεί υπόψη όταν είχαμε τις ακροάσεις των επιτρόπων. Εδώ εμείς μιλήσαμε για την ιδιαιτερότητα της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά δεν θεωρούμε ότι μας άκουσαν ή μας κατάλαβαν οι επίτροποι. Και αυτό μας ανησυχεί σε σχέση με την ανακοίνωση που θα βγάλει η Κομισιόν. Αλλά εντάξει, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις η ευαισθησία λαμβάνεται πολύ περισσότερο υπόψη λογικά από πλευρά Συμβουλίου. Όμως δεν είναι προφανές ότι η ατζέντα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου είναι και πολύ φιλόδοξη. Επομένως, καλό είναι εμείς να κάνουμε κάποιες συστάσεις, κάποιες υποδείξεις. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και ο Μίκαλ Γκάλερ και η Μαριαλένα Κοπά ε, θα μας υποστηρίξουν, ε, θα ετοιμάσουν την ετήσια έκθεση για την ΚΠΑ και θα είναι η πλατφόρμα για την παρουσίαση των θέσεών μας πριν το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Στο μεταξύ θα υποδεχθούμε κάποιους υπουργού Άμυνα, αλλά και κάποιους άλλους θεσμικούς παράγοντες. Και τώρα θα μετά από όλα αυτά θα αφήσω το λόγο στους επόμενους και φαντάζομαι θα εκτιμήσουν το ότι τους δίνω και λίγο χρόνο παραπάνω, λίγη πίστοση χρόνου.

Uh, Περνάμε στο δεύτερο σημείο της σημερινής διάταξης. Έταση της έκθεσης πρωτοβουλίας της κυρίας Γιαννάκου σχετικά με τις στρατιωτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές. Please. Έχουν κατατεθεί 104 τροπολογίες. Η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαΐου στην ΑΦΕΤ λόγο έχει η κυρία Γεννάκου για να μας παρουσιάσει τις θέσεις της επί των τροπολογιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, παρότι νομίζω ότι δεν, δεν ξέρω αν έχει και νόημα δηλαδή, διότι εδώ δεν υπάρχουν μέλη. Και ομολογώ ότι, εν πάση περιπτώσει. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που έκαναν ε, και ιδιαίτερα τους σκιώδεις συγητές γιατί είχαμε καλή συνεργασία μαζί τους. Το θέμα της έκθεσης βέβαια είναι τέτοιο που από τη φύση του είναι λογικό να υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις καθώς η άμυνα είναι ένας τομέας που κατεξοχήν βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα του κράτους και της ευθύνης κάθε χώρας και τα κράτη-μέλη είναι ιδιαίτερα διστακτικά για να παραχωρήσουν αρμοδιότητες σε ευρύτερα σχήματα. Ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω από την αρχή τα κύρια σημεία της έκθεσης γιατί είναι κάτι που έχουμε συζητήσει εκτενώς σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα θέλω να ενημερώσω ότι τελικά λόγω υπερβολικού φόρτου στην ατζέντα του Ιουλίου η έκθεση θα έρθει στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου παρουσία της κυρίας Άστον. Η αλλαγή αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα με την ύπατη εκπρόσωπο, εν ώψη μάλιστα του κρισίμου συμβουλίου ε, στα τέλη του 2013. <coughs> Τώρα, ως προς την έκθεση. Όπως είπατε, έχουμε 104 τροπολογίες. Μετά τη συνάντηση με τους κοιόδης συγητές των άλλων πολιτικών ομάδων, καταλήξαμε σε 5 συμβιβαστικές και 7 oral amendments. Για τις συμβιβαστικές, η συμβιβαστική τροπολογία 1 είναι ουσιαστικά ένα συνδυασμό από προσθήκε τη παραγράφου 1 και 2. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα, διότι οι προσθήκε είναι συμπληρωματικέ και βελτιώνουν το αρχικό κείμενο. Εξυπακούεται ότι έχουμε συζητήσει με του σκιώδη εισηγητές. Η συμβιβαστική 2 αναφέρεται στην παράγραφο 4 και αυτή είναι μια συλλογή από προσθήκες συμπληρωματικού χαρακτήρα. Η συμβιβαστική 3 στην αρχική παράγραφο 17 καλύπτει τις τροπολογίες 51 του κυρίου Νταμζόν και και την τροπολογία 52 της κυρίας Νικολάη. Ε, νομίζω ότι είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός καθώς ακόμα και ο αναθεωρημένος μηχανισμός Ατένα δεν λαμβάνει επαρκώς τις ιδιαιτερότητες των EU Battle Groups και πρέπει να προσαρμοστεί περαιτέρω προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό κοινών δαπανών διασφαλίζοντας επομένως το δικαιότερο επιμερισμό της επιβάρυνσης όταν έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η συμβαστική 4 αναφέρεται στην παράγραφο 19 και καλύπτει τις τροπολογίες 56 Πασκού, 57 Λίζεκ, 58 Γκάλερ Γιαννάκου, 59 Νταφ Ντανζόν. Ήξερα από την αρχή ότι πρότασή μου να προτείνω την έναρξη μιας συζήτησης σχετικά με την ανάθεση στην ύπατη εκπρόσωπο ορισμένων περιορισμένων εξουσιών όσο αφορά στην ανάπτυξη των EU Battle Groups για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα ήταν αμφιλεγόμενη και ίσως παρεξηγήσιμη. Νομίζω ότι ο συμβασμός λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές απόψεις και είναι ιδιαίτερα ισορροπημένος. Απλουστευμένες διαδικασίες για την ανάπτυξη των ομάδων μάχης είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, η συμβαστική 5 καλύπτει τις τροπολογίες 91 DAF, 92 λιζεκ 93-94 Μπασέσκου και αναφέρεται στη συνεργασία της ΥΠΑ της εκπροσώπου και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Τονίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη των υφισταμένων ήδη πλαισίων συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Κατόπιν συζήτηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων κύριο Μπρόκ και την εισηγήτρια της έκθεσης πρόοδου για την Τουρκία κυρία Όουμεν μου ζητήθηκε να κάνουμε μια προσθήκη στο τέλος της συμβαστικής αυτής η οποία θα αναφέρεται στην μη εφαρμογή από την Τουρκία των Berlin Plus Agreements. Ε, στην αρχή το θέμα είχε τεθεί ως μη κύρωση από την ε, Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση της απόφασης αυτής, αλλά η Γραμματεία με πληροφόρησε ότι δεν υπάρχει κύρωση, ούτε χρειάζονται κυρώσεις. Ε, η Τουρκία δεν επιτρέπει την εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα ότι ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ ισχύει ο κανόνας της ομοφωνίας. Η προσθήκη λοιπόν είναι η εξής. Στην τροπολογία 5, στο τέλος, starting from the Berlin Plus agreements, which Turkey will block their implementation. Αυτό είναι καλύτερο ε, και νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Βέβαια θέλω να έχω και την γνώμη των άλλων πολιτικών ομάδων επ' αυτού, γιατί αυτό ήρθε τελευταίο προχθές. Όσο αφορά στις προφορικές τροπολογίες, είναι κυρίως ενημέρωση κάποιων προσφάτων εξελίξεων, κάποιες επαναδιατυπώσεις, ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν από περισσότερες πολιτικές ομάδες. Ε, κυρία Πρόεδρε, είναι προφανές ότι πρέπει να εξετάσουμε τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των δεσμεύσεών της στη διεθνή ασφάλεια και στη διαχείριση κρίσεων. Η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας είναι βέβαια το ζητούμενο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται καλύτερος συντονισμός του αμυντικού σχεδιασμού οι συνέργειες που μπορούν να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να αποτελέσουν και τη λύση στα προβλήματα που επιβάλλει το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο. Δυστυχώς ως σήμερα δεν υπάρχει σαφής δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών για να αναπτυχθούν οι αναγκαίες ικανότητες αλλά και να ενεργοποιηθούν και να υποστηριχθούν οι υπάρχουσες δομές όπως είναι τα battle groups. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και να κάνουν ένα βήμα μπροστά στην κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Και γι' αυτό το λόγο η ύπατη εκπρόσωπος πρέπει να παρουσιάζει σαφείς προτάσεις. Η έκθεση δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα προς αυτήν την κατεύθυνση που είναι και φιλόδοξα και θα έλεγα και ρεαλιστικά. Θεωρώ ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα εν ώψη του κρισίμου Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και να απαιτήσουμε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και όχι απλά ευχολόγια και δηλώσεις καλών προθέσεων, διότι το σύστημα έχει κατηθυλωθεί στην ε, ουσία στα όσα ε, αποφασίστηκαν στην αρχή αυτής της δεκαετίας, η οποία είχε ήδη εκπνεύσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιαννάκου. Συμφωνώ απόλυτα με τις διαπιστώσεις σας ε, ότι χρειάζεται αναθεώρηση όλων των ε, δομών και αξιολόγησή τους γιατί ε, πηγαίνουν πολύ πίσω στην αρχή ε, της προηγούμενης δεκαετίας. θέλω εκ μέρους του σκιώδους συζητητή της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να σας διαβάσω την παρέμβασή του διότι δεν μπορούσε να είναι εδώ. Our shadow Κύριος Πάσκου, ε, λυπάται που δεν ήταν σε θέση να συμμετάσχει στη σημερινή συζήτηση. Ε, ε, μιλάει σε ένα διεθνές συνέδριο στη Ρουμανία και είχε δεχτεί αυτή την δέσμευση πολύ πριν να κανονιστεί αυτή η συνάντηση. Όμως συμμετείχε στην συνάντηση των σκιωδών με την εισηγήτρια και θέλω να παρουσιάσω τη θέση, της, τη θέση του τώρα. Όπως υπόθηκε σε προηγούμενες συζητήσεις, υποστηρίζουμε τη βασική ιδέα και ε, το σχέδιο της έκθεσης κυρίας Γεννάκου. Είναι επίκαιρη έκθεση με ουσιαστικές προτάσεις για την βελτίωση της ε, στρατιωτικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη του ε, επερχόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Οι τροπολογίες στην έκθεση, ως συνήθως, είναι επικύλες και σημαντικές. Υποστηρίζουμε τις τροπολογίες που προσθέτουν αξία στην ε, έκθεση. Η ομάδα μας απορρίπτει τις τροπολογίες που προσπαθούν να εξαλείψουν για διαφορετικούς ιδεολογικούς λόγους τις προτάσεις της έκθεσης για βελτίωση της ε, στρατηγικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υποστηρίζουμε φερειπίν την τροπολογία, ε, τις τροπολογίες που θέλουν να ακυρώσουν θετικά πράγματα που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες εκθέσεις. Υπάρχουν τρία σημεία που ο κύριος Πάσκου θα ήθελε να τονίσει. Πρώτον, συμφωνούμε με έναν ε, συμβιβασμό που συγκερνά τις απόψεις διαφορετικών πολιτικών ομάδων. Κάποιες ε, από τις τροπολογίες της ε, σκιώδους συγκήτριας υπάρχουν ήδη στο συμβιβασμό. Έχουμε ένα καλό παράδειγμα στο συμβιβασμό 4 που καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διερευνήσει τρόπους απλούστευσης των πολιτικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ούτω ώστε να γίνει πραγματικότητα η γρήγορη αντίδραση. Ε, η σκέψη για απλουστευμένες δικασίες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη μάχημων ομάδων για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα βασίζεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα έχουν προσυμφωνηθεί όπως ε, ζήτησαν και τα Ηνωμένα Έθνη. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του κ. Πάσκου, ε, μιλάει για την ανάγκη πλήρους προσέγγιση για την διαχείριση των κρίσεων, ε, ενσωματώντας διπλωματικές, οικονομικές εξελίξεις και, αν δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, στρατιωτικά μέσα. Ο σχεδόν συζητητή θέλει την ενίσχυση τη περιφερειακή διάσταση των μάχημων μονάδων, ούτω ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του. Μαζί με την εισηγήτρια, ο κ. Πάσχου ε, ζητάει αξιολόγηση της δημιουργίας μιας μόνιμης, ενός μόνιμου κέντρου ε, της ΚΠΑ ε, τέλος, ο κύριος Πάσκου θέλει να επαναλάβει την εκτίμηση της α, επικοδομητικής συνεργασίας που είχε με την κυρία Γιαννάκου για την σημαντική αυτή έκθεση. Η ομάδα μας θα υποστηρίξει όλα τα σημεία που προωθούν ε, πιο αποτελεσματική χρήση των υπαρχουσών ε, στρατιωτικών δομών και της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. of the Socialist Group, Mrs. Κλείνει το μικρόφωνο της Προέδρου. Αυτά ήταν τα σχόλια των σοσιαλιστών, κύριε Γιαννάκου. Θέλετε να απαντήσετε στα σχόλια του κύριου Γιαννά... Ε, Πάσκου. Ε, η συνεργασία μας με τον α, α, σκιώδη εισηγητή της Σοσιαλιστικής Ομάδος υπήρξε εξαιρετικά επικοδομητική. Α, ε, με είχε ειδοποιήσει προκαιρού ότι δεν θα μπορούσε να είναι σήμερα εδώ και ορισμένες από τις προτάσεις του είχαν ήδη ενταχθεί μέσα στην α, εισήγησή μου ακόμα πριν γίνουν οι διάφορες τροπολογίες. Ε, έχω την εντύπωση ότι ε, η έκθεση και με τη βοήθεια ε, των άλλων ομάδων αλλά κυρίως του κυρίου Πάσκου μπορεί να γίνει αποδεκτή σαν ένα, μια προσπάθεια να γίνουν πολύ συγκεκριμένα βήματα άσταση την οποία και εσείς οι ίδια περιγράψατε προηγουμένως αφενός και ταυτόχρονα δεν νομίζουμε ότι δημιουργεί ε, ή μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις ε, ως ε, έκθεση η οποία προτείνει υπερβολικά επαναστατικές αλλαγές. Όχι γιατί δεν θα ήθελα εγώ ως εισηγήτρια, αλλά γιατί καλό είναι και χρήσιμο αυτά που προτείνονται να μπορούν να γίνουν και να υποστηριχθούν από όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία όπως είπαμε και στην αρχή έχουν διάφορες επιφυλάξεις που προέρχονται πολλές φορές και από την ιστορικότητα ορισμένων πράξεων και πραγμάτων αλλά και κυρίως από το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό θεωρείται σκληρός πυρήνας του κράτους. Νομίζω ότι στην ψηφοφορία η οποία θα γίνει μέσα σε αυτή τη βδομάδα ε, θα μπορούμε να έχουμε ως αποτέλεσμα μια έκθεση ισορροπημένη. Εγώ θα στείλω την Τετάρτη σε όλους ε, τους ε, σκιώδεις εισηγητές τη δική μου πρόταση για την ψηφοφορία. Για το πώς Έχουν ήδη στα χέρια τους οι σκιώδεις εισηγητές τη σειρά των τροπολογιών, έτσι όπως εκτίθενται προς ψήφιση και θα στείλω και την δική μου πρόταση ε, για το πώς θα επιθυμούσα ή νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε και αυτό μπορεί να συνεκτιμηθεί και από τους άλλους και συζητητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γιαννάκου. Η, επαναλαμβάνω ότι είναι ψηφοφορία για τις 30 Μαΐου ε, και θα ήθελα να μεταφερθεί παρακαλώ σε όλους τους ευρωβουλευτές που είναι απόντες ότι λόγω της μεγάλης σημασίας αυτής της έκθεσης καλό είναι όλες οι πολιτικές ομάδες να ειδοποιήσουν για συμμετοχή στην ψηφοφορία γιατί τέτοιου είδου εκθέσει έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον τη Ένωση και η συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι ε, κομβική σημασία. Ιδίω και εν ώψη των ευρωεκλογών, όπου δεν είναι ωραίο σημαντικέ εκθέσει να περνούν με πολύ ε, μικρή συμμετοχή. Οπότε αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω και τη Γραμματεία να το φροντίσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, η επόμενη συνάντηση είναι για τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, 3.30 η ώρα το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνεδρία συλλήεται. Φαίνεται ότι είναι όλοι υπέρ. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. <laughs> Λοιπόν,